So good, afternoon, everybody. Sorry to keep you uh, waiting, but I had a meeting down at and the traffic's very bad. So, uh, Είναι πολύ φορτισμένη κυκλοφορία και γι' αυτό άργησα λιγάκι. Συγγνώμη. Θέλω να δω αν η κυρία Μπίλτ θα έρθει. Α, εσείς είστε λοιπόν η κυρία Κοράτσα Μπίλτ για το απόγευμα την, την, αντα, την αντικαθιστάτε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, όλοι είναι εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι. Και καλωσορίζω και όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Υπάρχει και ένα Άλλαξα μικρόφωνα, λέει ο πρόεδρος, γιατί χρησιμοποιώ κυρίως το αριστερό μου χέρι. Έχουμε λοιπόν ένα καινούριο newsletter για σας. Εάν κοιτάξατε τα δεδομένα του λιανικού τομέα και θέλατε να ενημερωθείτε για τη συζήτηση το απόγευμα. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν σημαντικά στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση και γι' αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα τις ε, συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες έχουν συζητήσει σκιώδεις προετοιμάζοντας την ψηφοφορία μας στις 5 Νοεμβρίου. Και χωρίς, να, για να μην μακρηγορώ δίνω το λόγο στον εισηγητή. Σε ευχαριστώ Μάλκομ. Θα είμαι σύντομος. Πιστεύω ότι μπορώ να είμαι σύντομο, σύντομος, διότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες κάθε συμβιβαστικής τροπολογίας. Είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συνάντηση στο Στρασβούργο την περισμένη εβδομάδα με τους κοιόδης εισηγητές και ορισμένες λεπτομέρειες ακόμα εκρεμούν. Μετά τη συζήτηση έκανε ορισμένες αλλαγές, ορισμένες τροποποίησεις και προσέθεσα και μερικές νέες τροπολογίες που αφορούν την υλοποίηση της νομοθεσίας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για της εσωτερικής αγοράς και κρεμούν ακόμα ορισμένες προτάσεις σε διάφορα σημεία. Αντί λοιπόν να συζητήσουμε μία προς μία, τις ε, ομαδοποιήσουμε ε, σε ένα νέο ε, συμβιβασμό που είναι ο πέντε η τροπολογία 5, συμβιβαστική θα με ενδιαφέρει να ακούσω από άλλα μέλη και τους κοιόδης εισηγητές αν αυτή η δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών ε, ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, την επισημητή κατεύθυνση και ε, πιστεύω ότι θα χειριστούμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες περισσότερο μέσω της γραπτής διαδικασίας, διότι την ερχόμενη εβδομάδα στο Ασβούργο έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας. Οπότε, όσα εκκρεμή ζητήματα ακόμα υπάρχουν, καλύτερα να τα λύσουμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. So, let's, uh, Ωραία. Λέω, ο Πρόεδρος, ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Μπόρισοφ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Ντεγιάνγκ, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κορέτσα Μπίλ θέλει να σας ευχαριστήσει για την επιτυχή συνεδρίαση και μου ζήτησε να σας ενημερώσω για τα βασικά θέματα. Πιστεύει ότι έχουμε μια καλή βάση εργασίας, αλλά πρέπει ακόμα να ασχοληθούμε με ορισμένα εκκρεμή ζητήματα. Πρώτον, στην ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να επιμείνουμε στην ε, σωστή υλοποίηση της νομοθεσίας ε, της εσωτερικής αγοράς. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που ο εισηγητής στις ε, ενημερωμένες, στις επικαιροποιημένες τροπολογίες έχει ενσωματώσει τις, τις προσεγγίσεις μας, τις ιδέες μας ή όποιε περιλαμβάνουν κυρίως θέματα διασυνοριακών, διασυνοριακής κυκλοφορίας. Δεύτερον, όπως συζητήσαμε στην ε, συνάντηση των ε, σκιωδών, το πρόγραμμα δράσης είναι ένα ζωντανό κείμενο και δεν χρειάζεται να ξαναξεκινήσει η συζήτηση από την Κομισιόν. Θα πρέπει τώρα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και να απευθυνθούμε στους ενδιαφερόμενους και τις τοπικές αρχές και να ζητήσουμε να προχωρήσουν περαιτέρω στο πρόγραμμα δράσης μέσα στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κανονισμών για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ε, ανθρώπων ε, προς τις, ε, και επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να επιτύχουμε μια καλύτερη ισορροπία για να δώσουμε περισσότερη ευθύνη σε αυτούς που ασχολούνται με την αηφορία, που είναι υπεύθυνοι για την αηφορία και να δώσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές για μικρά ε, καταστήματα μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τις ε, θεμητές ε, εμπορικές πρακτικές, η θέση μου είναι ξεκάθαρη δεν θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιό να προτείνει άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις ή κυρώσεις. Αυτό θα προκαταβάλει ε, την μελέτη αντικτύπου, αντικτύπων και θα περιορίσει τις διάφορες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα. Εδώ έχουμε πετύχει μια ιστορική συμφωνία επί τη βάση των βέλτιστων πρακτικών και επί τη βάση των μηχανισμών υλοποίησης ε, των προτάσεων ε, από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Πάνω από 450 ενδιαφερόμενοι έχουν ε, δεσμευτεί στο να ε, υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό πρέπει να πιέσουμε για την ταχύτερη εφαρμογή ε, και να, να παρακολουθούμε την εξέλιξη τακτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες πρόσβασης και η νομοθεσία τώρα θα πρέπει απλώς να συμπληρώνει το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο. Ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους τους συνάδελφους που συνεργάστηκαν επικοδομητικά και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του εισηγητή. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγιόγκα για την καλή δουλειά που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Ελοποιήσαμε μία συνεδρίαση με αυτόν και τους Σκιώδης και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις συμβιβαστικές προτάσεις τις αρχικές. Ο εισηγητής ήδη έχει συμπεριλάβει τις ανησυχίες της ομάδας μου που εξέφρασα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης και τις έχει συμπεριλάβει στο κείμενο. Θα ήθελα να αναφέρω τις πέντε συμβαστικές τροπολογίες που θεωρώ ότι είναι απαραίτητες και σημαντικές για την ομάδα μου υπαρχημών 4 για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, συμβιβαστική υπαριθμών 5, σχετικά με τη σημασία των διοικητικών εμποδίων που εμποδίζουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι' αυτό η ομάδα μου προτιμά την αναδιατύπωση που προτείνει ο εισηγητή για το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 5 όπου συμπεριλαμβάνει την πρότασή μας, συμβαστική τροπολογία 10. Εδώ χαιρόμαστε που παραμένει η αναφορά στους παραγωγούς ε, και των τρίτων χωρών, ε, αλλά θέλουμε να συμπεριληφθούν ε, και οι εργαζόμενοι. Το σημείο 11 είναι σημείο κλειδί για την ομάδα μου. Χαιρετίζουμε που παραμένει η έκκληση στην Κομισιόν για να θεωρηθούν τα πρακτικά αποτελέσματα της εθελοντικής πρωτοβουλίας συμπεριλαμβανομένων και της υλοποίησης των βελτιστών πρακτικών μετά από ένα χρόνο της και να αξιολογηθεί η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων. Θέλω να τονίσω τη μεγάλη δουλειά που έγινε για να τεθεί σε εφαρμογή εξουσία πρωτοβουλία. Αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να αξιολογήσουμε τα πιθανά προβλήματα του συστήματος και να τα διορθώσουμε έτσι λοιπόν υπολογία υπερθυμών 13 για τις συνθήκες εργασίας και την αποζημίωση των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων ε, διανομής. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην 4α σε σχέση με την εθνική ε, φορολογική και εμπορική νομοθεσία που θίγουν συγκεκριμένα μοντέλα επιχειρηματικά και διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Εμείς, όπως είπαμε και στη συνεδρία των σκιονοδών εισηγητών, δεν υποστηρίζει την πρόταση αυτή γιατί θεωρούμε ότι αυτή αυτό είναι ο στόχο αυτή τη ζήτηση, και σε σχέση με τη νέα πρωτοβουλία για τη νέα παράγραφο 5α η ομάδα μου συμφωνεί με την αναγκαιότητα να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη το πόσο σημαντικό είναι να μεταφέρουν σωστά στο ιστορικό τους δίκαιο την ομοθεσία και να απαιτήσουν μια πολιτική μηδενική ανοχή για τα κράτη που δεν εφαρμόζουν όπω πρέπει του κανόνε τη εσωτερική αγορά. Ωστόσο θεωρώ ότι η παράγραφος ε, είναι υπερβολικά μακροσκελή. και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγιόν για την εξαιρετική δουλειά του στην προετοιμασία τη εκθέση αυτή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Mr. Lückegaard is next. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συγγετή για την ε, καλή συνάντηση την περασμένη εβδομάδα. Κάναμε πρόοδο και νομίζω ότι τα περισσότερα από τα θέματα συζητήθηκαν σοβαρά και Τώρα βλέπουμε μια σοβαρή απόπειρα να σημειωθεί πρόοδος. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο εισηγητής μέχρι τώρα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια σχόλια για τις, ε, για τις τροπολογίες χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Οι πρώτες έξι τροπολογίες, κατά την άποψή μας, είναι εντάξει, αλλά αρχίζουν τα προβλήματα στην υπαριθμό 7. Εξακολουθεί να μην είναι σαφές για μένα Ποιο είναι ο σκοπός της τροπολογίας 7. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Με πάρα πολλά λόγια περιγράφεται κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να περιγραφούμε τόσο πολλά λόγια. Θέλω να το ξανασυζητήσουμε για την 8, για τα shopping centers, για τα εμπορικά κέντρα. Εδώ συμφωνώ με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ ότι δεν ε, ε, μπορούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και δεν ξέρω αν είναι δυνατό να συμφωνήσουν και άλλες ομάδες. Γιατί επί της αρχής νομίζω ότι είναι κάπως παράξενο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό έτσι όπως περιγράφεται εδώ αλλά εξακολουθούμε να είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Όμως μέχρι τώρα δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η προσέγγιση αυτής της τροπολογίας. Ε, αν διορθωθεί θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για την ε, υπαριθμόν 9. Έχω μια ερώτηση. Φυσικά έχει γίνει πρόοδος ε, για κάποια συνοσημασία θέματα. Εδώ καλωσορίζουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 9. Σε σχέση με το δεύτερο τμήμα δηλαδή την ε, απαγόρευση για το μηχανισμό καθορισμού των τιμών στα συστήματα franchise. Μου ακούγεται κάπως περίεργη αυτή η διατύπωση. Ίσως θα μπορούσαμε να προτείνουμε να χωριστεί αυτή η τροπολογία στα δύο. Θα το ξανασυζητήσουμε. Η 10 εντάξει. Σε ό,τι αφορά την 11. Και εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση για το τελευταίο τμήμα, τελευταία φράση. Όταν αναφερόμαστε σε αυτούς τους επιπρόσθετους ανεξάρτητους μηχανισμούς επιβολής, τι εννοούμε εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε ξεκάθαρα γιατί πράγμα μιλάμε για να δούμε αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Θέλουμε μια σαφή απάντηση και αν είναι αποδεκτή θα μπορούσαμε να την υποστηρίξουμε όσο έχει. Οι 12 και 13 μας βρίσκουν αντίθετους, αλλά δεν θα εκπλήξει αυτό τον εισηγητή. Αλλά συνολικά νομίζω ότι είναι καλή δουλειά σας μέχρι τώρα. Και όπως είπα, είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω συζητήσεις για τις τροπολογίες που ανέφερε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούλα. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι Λυπάμαι και συμφωνώ με πολλά που είπε ο συνάδελφός μου, ε, δεν βοηθούμε ε, το λιανικό εμπόριο εάν δεν κατονομάσουμε τα προβλήματα για να τα ξεπεράσουν. Ε, το μόνο που αναφέρεται το άρθρο 12, παράγραφος 12, λέει ότι η Κομισιόν η, ε, παρακαλεί την Κομισιόν να εξετάσει εάν ε, μπορεί να ε, χειριστεί καλύτερα και να απαντήσει καλύτερα στα παράπονα. Εάν αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει, να ξεφύγει από τον έλεγχο και να ασκείται πλέον τεράστια πίεση, έχουμε χάσει ε, ε, το δρόμο μας. Ε, πρέπει να απευθυνθούμε πλέον στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διχογνωμίες, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να τις επιλύσουμε. Οι τροπολογίες 10, 11, 12, 13 είναι οι ουσιαστικές, διότι απαντούν, ανταποκρίνονται και στα υπάρχοντα προβλήματα. Όσον αφορά τώρα την ε, ε, εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, συμφωνώ ότι δεν θέλουμε να αυξήσουμε το, το νομοθετικό βάρος, αλλά ε, πώς θα πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες εφαρμογής, επιβολής της νομοθετικής των νομοθετικών κανονισμών και του πλαισίου αυτού. Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να είναι σε λούσια η εφαρμογή του πλαισίου αυτού. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο παρακολούθησης και υλοποίησης. Με ποια μορφή. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να βοηθήσει ο διαμεσολαβητής να επιλύσει τέτοια προβλήματα. Τα οποία προβλήματα, μην κρυβόμαστε, ε, αφορούν ε, διαφορετικούς τομείς στο όλο λιανικό εμπόριο. Δεν έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα, πολλών τα συμφέροντα είναι αντικρούμενα και πολλοί επισημούν να έχουν ένα μηχανισμό ε, Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, μπορούμε να, εφαρμόσουμε καλύτερα και να παρακολουθήσουμε, να υποπτεύσουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι οι προτάσεις της εισηγήτριας είναι ε, θα αποτελέσουν μια σωστή βάση του εισηγητή, μια σωστή βάση συμβιβασμού και θα υποστηρίξουμε όπου μπορούμε. Well, so I'm... Λοιπόν, θα συμφωνήσω ως σκιώδης εισηγητής. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι στη συνάντηση των σκιωδών πέρσι, ε, την περιορισμένη εβδομάδα, συγγνώμη. Αλλά ε, κάποιος με εκπροσώπησε, ξέρω ότι εξετάσατε τις συμβιβαστικές τρυπολογίες, μπορούμε να στηρίξουμε πολλές από αυτές, το έχουμε ήδη πει. Για να προχωρήσουμε λοιπόν σήμερα, να τονίσω μόνο κάποια προβληματικά σημεία, τα οποία είναι πολύ παρεμφερή με αυτά που επεσήμενε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και ο κύριος Λιφκιακάρ. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο. Για τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Πώς παρουσιάζονται αυτά τα ζητήματα Κάθε κράτο μέλο έχει ξεχωριστό θέμα και έχει και διαφορετική νομοθεσία για να τα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαι πεπισμένο ότι είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το καλύτερο είναι να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το θέμα. Δεν το πιστεύω αυτό. Η Επιτροπή έχει πολλά στοιχεία και έχει βαθμολόγιο για την καταναλωτική συμπεριφορά και την αγοραστική συμπεριφορά αλλά άλλο θέμα είναι αυτό και άλλο θέμα ε, το θέμα της τιμολόγησης. Η δική μας επιτροπή ίσως δεν θα πρέπει να ασχοληθεί τόσο με αυτό. Γιατί δεν είναι τόσο θέμα εναρμόνισης. Και από εκεί και πέρα, μας ε, έχει εφιστήσει την προσοχή κάποιος και δεν μας εκπλήσει αυτό, γιατί πολλοί ενδιαφέρονται, στο ότι εδώ υπάρχει μια δήλωση και λέμε ότι τα εμπορικά κέντρα συνήθως έχουν υψηλότερες τιμές από ότι τα απλά καταστήματα, τα ανεξάρτητα. Κάποιοι όμως θεωρούν το αντίθετο. Εμείς δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε αυτό ή το αντίθετό του ανεξάρτητα και αντικειμενικά. Να μην κάνουμε λοιπόν τέτοιους ισχυρισμούς οι οποίοι είναι αβάσιμοι. και ίσως θα πρέπει να ε, προτείνουμε στον εισηγητή διατύπωση για να το τροποποιήσει αυτό. Τώρα, για τις συμβαστικές τροπολογίες 11 και 12, στις οποίες αναφέρθηκαν διάφοροι συνάδελφοι. Θα πρέπει να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά περιλαμβάνονταν στις αρχικές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μηχανισμούς θέση σε ισχύ σε θελούσια βάση σε διάφορα κράτη-μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα μηχανισμό που βασίζεται σε καταστατικό χάρτη, σε καταστατικό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες εξελίξεις παντού. Άρα εδώ τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να συλλέξουμε στοιχεία και να παρακολουθούμε τις νέες αυτές πρωτοβουλίες, να δούμε τι ε, αποτέλεσμα θα φέρουν στην πράξη, ποιον αντίκτυπο θα έχουν στην πράξη. Και θα πρέπει να ε, δούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ενιαία αγορά μέσω των διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής και να έχουμε ρυθμίσεις και διευθετήσεις κατά της κατάχρησης ε, δεσπόζουσας θέσεις. Κατά των καταχρήσεων μάλλον γενικότερα. Ίσως θα πρέπει να παρέμβουμε για την θέσπιση μηχανισμών διαιτησίας. Ωστόσο, η δική μου άποψη και της ομάδας πιστεύω ότι δεν είναι εξουσία του, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κάθε χώρα έχει διαφορετικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Δεν θα πρέπει να προσφεύγουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εάν λοιπόν οι δύο αυτές τροπολογίες μπορέσουν να αντικατοπτρίσουν καλύτερα την κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή με αυτά τα εθελούσια συστήματα, και αν δείξουν με καλύτερο τρόπο ποια είναι η πρόθεση και πώς θα προχωρήσουμε, τότε θα τίνουμε περισσότερο να τις υποστηρίξουμε. Από εκεί και πέρα, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τον κύριο Λίκεργαρντ, με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ για το θέμα της τιμολόγησης, για την απαγόρευση των πωλήσεων κάτω του κόστους και για διάφορα άλλα, τα οποία ίσως ε, Χρειάζεται να παρεύουμε χωρίς όμως να παρεύουμε και υπερβολικά στην αγορά. Ε, επιπλέον, οι κάθετοι περιορισμοί στα συστήματα εφοδιασμού, ε, όλα αυτά που έχουν να, ε, να κάνουν πολύ με τις αλλαγές στη διανομή των εμπορικών σημάτων είναι κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και η Κομισιόν μας ζητά την άποψή μας για όλα αυτά. Θα πρέπει δηλαδή κάπως να αναφερθούν ρητός όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν τα καλύπτει αυτά η τροπολογία 61. Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα ψηφιστεί συμπληρωματικά με κάποιες από τις άλλες τροπολογίες που είναι δικές του. Αυτά γενικώ θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ως προς την δέσμη των τροπολογιών που προτείνεται. Νομίζω ότι αν δουλέψουμε λίγο παραπάνω θα έχουμε μια εξαιρετικά πολύτιμη και χρήσιμη έκθεση. Θα προχωρήσουμε και θα έχουμε καλύτερες μελλοντικέ δράσεις, θα κατανοήσουμε καλύτερα και θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ε, όπου θα ενισχύουμε τη λιανική και θα εστιάζουμε ε, στον καταναλωτή. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Είναι και η Κομισιόν εδώ. Θέλει να σχολιάσει παρακαλώ. Όχι. Όχι σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστούμε. Καλώς. Καλό λοιπόν τον Τένις να μας συνοψίσει το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι σκιώδεις εισηγητές αλλά και όσοι τους εκπροσώπησαν για τα μετέφεραν τα σχόλιά τους ε, έκανα πολύ καλή δουλειά και τους ευχαριστώ πολύ. Κάποιοι είναι πιο ευέλικτοι από κάποιους άλλους σε ορισμένα ζητήματα. Μία από τις διαφορές που έχουμε με τους φιλελεύθερους ως προς τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8 είναι η εξής. Μίλησα, ε, διάβασα στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν την απαγόρευση του τέστην για τις οικονομικές ανάγκες. Και αυτό θα είναι μεγάλη πρόκληση για την Κομισιόν τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να δουν πώς τον εφαρμόζουν αυτή την νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό το εξής. Βεβαίως δεν πρέπει να ορίσουμε τις οικονομικές ανάγκες, αλλά θα πρέπει να αναφερθούμε ε, στην ανάγκη ύπαρξης μιας συγκεκριμένης πολιτικής, κάποιου σχεδιασμού τέλος πάντων από τις περιφερειακές και κεντρικές αρχές. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί αυτό να πλήξει υπερβολικά τα καταστήματα στις μεγάλες εμπορικές οδούς, ε, με το να εγκρίνει ο Δήμος τη την δημιουργία άλλου ενός, άλλου ενός εμπορικού κέντρου έξω από το κέντρο της πόλης, Αυτό δεν έχει σχέση με τις οικονομικές ανάγκες. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στο δικαίωμα των κρατών μελών και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης να δίνουν τέτοιες άδειες. Ε, βεβαιώσουμε ότι δεν θα παρέμβουμε στο Economic Needs Testing. Και είναι κάτι που φάνηκε και με τις τελευταίες συμβιβαστικές τροπολογίες ότι κανένα νομοθέτημα δεν θα πρέπει να δημιουργεί διακρίσεις. Ωστόσο, η τοπική αυτοδιοίκηση ή η κεντρική κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε κάποιο είδου σχεδιασμό. Έτσι δεν είναι. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει η διατύπωση να είναι λιγότερο ευέλικτη και στρέφουμε και στην τροπολογία υπαριθμών 7 για τα ανεξάρτητα σημεία ε, πώλησης, λιανικής πώλησης. Έχω μιλήσει με πολλούς εκπροσώπους του κλάδου και μου λένε ότι πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρητός αναγνωρίζει στο πλαίσιο της Λιανικής τη θέση των ανεξάρτητων λιανοπολιτών. Δεν νομίζω ότι πρέπει λοιπόν Ένα συμβιβασμό πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτό που μπορεί να γίνει αποδεκτό στι περισσότερε πολιτικέ ομάδε. Όλοι πρέπει να κινηθούμε, να αλλάξουμε το έδαφος. Καλό λοιπόν όλες τις ομάδες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τις τροπολογίες. Όπου είναι αυτό εφικτό, σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Αυτό πιστεύω. Και τέλος. Ε, Μια, ένα τελικό σχόλιο, σχόλιο για αυτό που είπε ο Μάλκομ για τα franchise. Είναι η τροπολογία υπαριθμών 9, τα ε, δικαιώματα ε, δικαιόχρησης. Μιλούμε για την τροπολογία του ECR και του Malcolm Harbour, όμως λέει και διαβάζω καλή η Κομισιόν και κρατημένοι να διασφαλίσουν ότι η απαλλαγή σε μπλόκο όλων αυτών ισχύει και εφαρμόζεται σωστά. Και το πρόβλημα των ε, αυτών που λαμβάνουν τη δικαιόχρηση είναι ότι ε, εάν αλλάξει αυτό θα πρέπει να είναι για να τοποθετηθούν εκείνοι καλύτερα. Δηλαδή το ECR λέει ότι το κείμενο είναι μια χαρά έτσι όπως έχει, δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί και ότι θα πρέπει να το αφήσουμε ως έχει. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλη αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό δεν το έβαλα. Να συμφωνήσουμε στη γενική ιδέα και να μην διευκρινίσουμε εάν θα ε, τροποποιηθεί ή το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί σωστά όλο αυτό το πράγμα. Μπορούμε να βάλουμε μια επίσημη αναθεώρηση. Αυτό καλύπτει όλους νομίζω. Καλό λοιπόν όλους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι στη διατύπωση που προτείνουν, να μου τα στείλουν αυτά με email και θα παρουσιάσω τελική εκδοχή των συμβιβαστικών τροπολογιών και τότε θα αποφασίσουμε αν θα συνεδριάσουμε για να τις ψηφίσουμε ή αν κάποιες από τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις αφήσουμε εκτός αφού δεν υπάρχει συνένεση. Ο Πρόεδρος. Ναι, οπωσδήποτε. Πιστεύω θα ανταποκριθώ σε αυτή την πρόσκληση γιατί από σήμερα μέχρι τις 5 Νοεμβρίου πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συντάξουμε μια εξαιρετικά καλή έκθεση που θα τύχει μεγάλη ευρεία υποστήριξης. Σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά για όλη σου την προσπάθεια. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Η είναι ο Ρόμπερτ Ροσφόρ και ε, τον συγχαίρω για την ε, ηγεσία που έχει δείξει στα θέματα του, των καταναλωτών, του καταναλωτισμού, ε, διότι επιτύχαμε μία συμφωνία και μια που δεν ήσουν παρόν στην αρχή της συνεδρίαση, θέλω να σε ευχαριστήσω τώρα. Έχουμε λοιπόν μία καινούργια έκθεση ε, που μας υπέβαλες για την εφαρμογή της οδηγίας για τις ΑΘΕΠ, αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και πάλι είναι παρούσα η Επιτροπή, θέλει κάποιος να λάβει το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής, ο κύριος Γκρέφκο. Ο κύριος Γκρέκο. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει και δύο λόγια για την προσέγγιση της Γενικής Διεύθυνσης ε, Δικαιοσύνης ε, μετά από την παρέμβαση των μελών. Η κυρία Ρούλε και εγώ θα συμβάλλουμε στη συζήτηση μετά, αλλά δίνω καταρχάς το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε βρεθεί μία φορά για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Έχετε λάβει λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι την πρώτη μου πρόταση έκθεσης και θα προσπαθήσω να σας την παρουσιάσω επιγραμματικά. Και με μεγάλη περιέργεια θα περιμένω τις αντιδράσεις σας και τις προτάσεις σας για συμπλήρωση και τροποποίηση του κειμένου αυτού. Τρία είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό περί του οποίου πρόκειται είναι η αξιολόγηση της, εφαρμογή, της, της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τρία ερωτήματα θύνεται, τίθενται λοιπόν. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το κείμενο της οδηγίας κάθε αυτό πρώτον. Δεύτερον, ποια είναι η γνώμη μας για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής και τρίτον, πώς θα καταφέρουμε έτσι ώστε οι καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το κείμενο, να, έχουμε, ε, ε, να έχουν εύκολα, γρήγορα αποτελεσματικά μέσα στα οποία να προσφύγουν, ούτως ώστε να υλοποιηθεί ο σκοπός. Δεν προτείνω έτσι όπως έχει η κατάσταση αυτή μεγάλη τροποποίηση του κειμένου της οδηγίας. Θεωρώ ότι το κείμενο είναι καλό, ότι λειτουργεί καλά η οδηγία και ότι μια αναθεώρηση εφόλης της ύλη δεν θα ήταν και το πιο σκόπιμο. Άλλωστε είναι μια οδηγία μέγιστης εναρμόνισης η οποία βασίζεται στον μαύρο κατάλογο των καταχρηστικών πρακτικών. Ωστόσο, η οδηγία μέγιστης εναρμόνισης, εκτός από τον κατάλογο αυτό, προβλέπει και τη δυνατότητα αξιολόγησης κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη. Αξιολόγησης αυτών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αθέμητοι ως αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ακόμα και αν δεν βρίσκονται σε αυτόν τον μαύρο κατάλογο, σε αυτή τη μαύρη λίστα. Δεν προτείνω λοιπόν μεγάλες τροποποιήσεις ουσιαστικές, Θεωρώ ότι το κείμενο πρέπει να διατηρηθεί ως έχει προς το παρόν και αυτό δεν εμποδίζει βεβαίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να, δημοσιεύει, να δημοσιεύει τη μαύρη λίστα με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές έτσι όπως τις παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη για λόγους καθαρά ενδεικτικούς έτσι ώστε να δούμε στο μέλλον πώς θα προσαρμόσουμε κατάλογα, κατάλληλα τη λίστα του παραρτήματος. Είναι μια συνεχή διαδικασία απογραφής, ωστόσο έτσι όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί αυτό το παράρτημα αυτό τώρα. Από εκεί και πέρα η οδηγία θα επεκταθεί, θα επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή της, εφαρμογής της δηλαδή στο business to consumer επίσης, όχι μόνο αλλά και όχι μόνο στο B2C, business to consumer, αλλά και στο B2B, στο, μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουμε την περιβόητη απάτη των τηλεφωνικών καταλόγων με τους αριθμούς ε, τους τηλεφωνικούς και τα ονόματα. Τη γνωρίζετε όλοι, έχει συζητηθεί το θέμα αυτό. Δεν νομίζω, και με ενδιαφέρει να μάθω και τη δική σας άποψη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν μπορούν να το κάνουν από, μόνοι, μόνα τους και μπορούν να το αποφασίσουν. Τέσσερις χώρες σήμερα το έχουν ήδη κάνει άλλωστε. Αυτό καταρχάς. Δεύτερον, το πώς θα εφαρμοστεί το κείμενο. Είναι σημαντικό. Θα ήθελα, και το λέω στην έκθεσή μου, να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες. Πρέπει να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και θα πρέπει να ε, παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία στα κράτη-μέλη και αν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται θα πρέπει η Κομισιόν να παρεμβαίνει δραστικά ε, να εγκαλεί τα κράτη που υπονομεύουν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Άλλωστε, ε, το τελευταίο στάδιο της μέγιστης εναρμόνισης έχει ξεκινήσει εδώ και μόλις λίγους μήνες. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι εθνικές αρχές, οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή και δεσμεύτηκε η Κομισιόν μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς να εξετάσει σε βάθος το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την προστασία των καταναλωτών και ενθαρρύνω την Κομισιόν να φέρει σε πέρα στο έργο αυτό, πόσο μάλλον αφού έχουμε αυτές τις επιχειρήσεις σκούπα που έχουν γίνει σε άλλους τομείς και που αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμες. Πρέπει να εντοπιστούν, να καταγγελθούν και να τιμωρηθούν, να υπάρξουν κυρώσεις για όλες αυτές τις πρακτικές και επιμένουμε στις κυρώσεις, διότι σαφέστατα σε ορισμένες καταστάσεις και σε ορισμένες χώρες μέλη οι κυρώσεις δεν είναι πραγματικά αποτρεπτικές. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, να μην αντικαθιστούμε τη δικαστική εξουσία, αλλά να πούμε ξεκάθαρα ποια κατεύθυνση θέλουμε να δώσουμε. Δεν θα πρέπει να μπορεί κανείς να αξιοποιήσει μια αθέμητη πρακτική. Δηλαδή οι κυρώσεις ποτέ δεν πρέπει να είναι κατώτερες από το κέρδος που αποκομίζει αυτός που προσφεύγει στην αθέμητη εμπορική πρακτική. Κάποιος που ε, ε, εφαρμόζει μια αθέμητη εμπορική πρακτική, αν ξέρει ότι αν πιαστεί αυτό που θα κληθεί να καταβάλει είναι πολύ λιγότερο από αυτό που θα κερδίσει, αυτό δεν είναι κίνητρο για να μην την κάνει αυτή την πρακτική. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα εργαλεία, τα μέσα, αυτά καθεαυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι δύο. Το έγγραφο προς ανατολισμού που συνοδεύει την εφαρμογή της οδηγίας και η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις καταστάσεις ε, που δίνουν λαβή για θέμητες εμπορικές πρακτικές. Καλό την ε, Κομισιόν να αναθεωρήσει το έγγραφο Ανατολισμού μέχρι τα τέλη του 2014 για να απεικονίζει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και ως προς τη βάση δεδομένων ξέρω ότι ζητώ κάτι πολύ, που είναι βαρύ ενδεχομένως, αλλά είναι μια βασή δεδομένων στα αγγλικά. Και αν θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν και να τη συμβουλευθούν και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες δηλαδή, θα πρέπει αν το επιθυμούμε αυτό σιγά-σιγά και σταδιακά να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεταφραστεί σταδιακά και σε άλλε γλώσσε της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βάση αυτή των δεδομένων. Θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν μέσα ένδικα προσφυγής γρήγορα αποτελεσματικά, χρήσιμα και θα πρέπει εμείς να τονίσουμε αυτή την ανάγκη, άλλωστε έτσι θα δείξουμε τι δουλειά έχουμε κάνει τα προηγούμενα εξάμηνα και τους προηγούμενους μήνες. Πρώτον, θα δείξουμε την σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, αλλά και για τους τρόπους εξοδικαστικής επίλυσης ε, συγκρούσεων διαδικτυακών με τη δουλειά της Κομισιόν αλλά και με το δικό μας προβληματισμό στη δική μας Επιτροπή ε, σκεφτόμαστε σιγά σιγά η Ένωση να φτάσει σε ε, συλλογικά μέσα προσφυγής που θα σέβονται τα συμφέροντα όλων των μερών. Άλλωστε, στον τομέα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη ε, γρήγορα να αποκτήσουμε μηχανισμό για συλλογικές προσφυγές. Δεν ξεχνώ τις οργανώσεις των καταναλωτών που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ούτε ξεχνώ τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και σας υπενθυμίζω τις ε, τρεις βασικές ιδέες της έκθεσής μου. Πρώτον, να μην τροποποιηθεί σημαντικά το κείμενο της οδηγίας. Δεύτερον, να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να βοηθήσουμε την Κομισιόν να βελτιώσει την εφαρμογή της οδηγίας. Και τρίτον, να έχουμε ε, προσβάσιμες οικονομικά ε, προσβάσιμα οικονομικά, αποτελεσματικά και γρήγορα μέσα προσφυγής. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πλήρη παρουσίαση των θεμάτων αυτών. Ε, να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους, ο κύριος Μπόρισεφ καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες Σεγητά. Σας ευχαριστώ για το επικοδομητικό σας ε, έργο και αν θέλουμε να έχουμε μία ενή αγορά θα πρέπει να προστατεύουμε τους καταναλωτές σε όλο αυτό το σύστημα. Θέλω κάποια σημεία να αναφέρω και θα μιλήσω τη μητρική μου. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιτείνουμε το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, ούτε χρειάζονται αλλαγέ ή τουλάχιστον μεγάλες ε, τροποποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι η εφαρμογή της οδηγίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ορισμένες ε, χώρες δεν εφαρμόζεται πλήρως. Επομένως, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Και η Κομισιόν όχι μόνο θα έπρεπε να παρακολουθεί τη διαδικασία της εφαρμογής, αλλά θα έπρεπε και να λαμβάνει προληπτική δράση και να παρέχει υποστήριξη έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις χώρες, οι χώρες στην οδηγία το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα, πιστεύω πως πρέπει να είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα οι κυρώσεις. Θα πρέπει να δοθεί εστίαση στην πρόληψη των καταχρηστικών πρακτικών οι οποίες δεν σέβονται τα συμφέροντα των καταναλωτών. Επίσης και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή τη μαύρη λίστα, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω. Φυσικά θα πρέπει να είναι αντικείμενο αξιολόγηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί γνωρίζουμε πως οι έμποροι, οι εμπορευόμενοι πάντοτε θα προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να ανακαλύψουν παραθυράκια. Και επίσης πιστεύω πως οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα Φυσικά θα πρέπει αυτό να γίνεται και σε προληπτικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ανυπομονώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενη ομιλήτρια, ευχαριστώ. Βρίσκομαι σε μια λεπτή θέση, γιατί δεν υπάρχει διερμηνία για μένα εδώ στην Επιτροπή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μεταφράσω την ομιλία μου στα αγγλικά. Θα προσπαθήσω να βάλω το δυνατά μου. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ροσφόρ για το σχέδιο της έκθεσης. Είναι καλό το κείμενο και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε από αυτού. Τώρα για ορισμένα από τα θέματα εδώ θα συμφωνούσα ότι η τρέχουσα νομοθεσία που υπάρχει για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, είναι αρκετά καλή και καλύπτει τις πιο προβληματικές πρακτικές. Επίσης συμφωνώ πώς θα πρέπει να αντιδικοποιήσουμε την επιβολή της νομοθεσίας και στο εσωτερικό των κρατών μελών, αλλά πρέπει να ενδυναμώσουμε και τη συνεργασία στις διασυνοριακές καταστάσεις. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξω τις ε, κρατικές αρχές ή τα κρατικά όργανα στις ελεγχτικές τους δραστηριότητες ό,τι αφορά την επιβολή του νόμου, αλλά επίσης θα ήθελα να υπάρχει και ένας ε, ρόλος των οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών. Αυτό δεν το βρήκα στο κείμενο, στο σχέδιο κειμένο, αλλά χαίρομαι πολύ που τα αναφέρατε στα εισαγωγικά σας σχόλια. Σε ό,τι αφορά τώρα στη συνεργασία, νομίζω ότι πρέπει να καλωσορίσουμε τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε από την Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή για την αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία των καταναλωτών και τη συνεργασία. Νομίζω ότι από εκεί μπορούμε να έχουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι καθώς έχουμε όλο ένα και πιο συνδεδεμένη εσωτερική αγορά και όλο ένα και περισσότερες διασυνοριακές και επιγραμμικές συναλλαγές, αυτό σημαίνει ότι τα μεμονωμένα όργανα επιβολής του νόμου είναι λιγότερο αποτελεσματικά στο να καταπολεμήσουν τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε πρακτικές ε, που βλέπουμε σε κάποιες εταιρείες που λειτουργούν διασυνοριακά. Επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά την επιβολή του νόμου μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό με οδηγεί στην εξή ιδέα. Αν έχουμε ένα ορμονισμένο νομοθέτημα για την προστασία των καταναλωτών, τότε θα πρέπει σοβαρά να σκεφτούμε την έννοια και της επιβολής αυτής της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τις τρίτες χώρες, νομίζω ότι καλή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες συναλλαγές στο διαδίκτυο, δεν ε, υπάρχει ίχνος ε, για το ποιος κάνει τη συναλλαγή και είναι ο domain εδρεύει σε μια τρίτη χώρα, τότε δεν υπάρχει καμία δίωξη και επιβολή κυρώσεων. Επίσης συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι προληπτικές και αποτρεπτικές οι κυρώσεις, όπως δηλώνεται στην οδηγία. Όμως ε, η εφαρμογή, επιβολή της νομοθεσίας είναι προβληματική. Δηλαδή, αν ένας φορέας επιβάλλει ένα τέλος ή μια κύρωση ή ένα πρόστιμο, δεν έχει κανένα feedback για το αν πληρώθηκε το πρόστιμο αυτό. από τον παραβάτη. Άλλες παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με τις κατευθυντήρες γραμμές κομισιών που συνοδεύουν την οδηγία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ανταλλαγής των πρακτικών μεταξύ της κομισιών και των φορέων επιβολής του νόμου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει για να βελτιώσουμε το έργο των οργανισμών αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα βελτίωσης εδώ και το τελευταίο μου σημείο έχει να κάνει με αποτελεσματικά και γρήγορα μέσα για τους καταναλωτές, όπως παραδείγματο χάρη η εναλλακτική επίλυση διαφορών, έτσι ώστε να μην καθυστερεί η εφαρμογή του νόμου. Και τέλος ελπίζω ότι με την έκθεση αυτή θα απευθύνουμε έκκληση για να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση για τη συλλογική προσφυγή. Σας ευχαριστώ. Ίσως να μην ήμουν πολύ ακριβή στην ορολογία, αλλά ανυπομονώ να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους σκιώδεις επί των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρούλε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Θερμά, γιατί και εγώ είχα αμφιβολία στην αρχή αν το χρειαζόμαστε αυτό ή όχι, αλλά πιστεύω τα επιχειρήματά σας είναι πολύ πιστικά και με πήρατε με το μέρος σας. Γι' αυτό συμφωνώ μαζί σας να μην γίνει αναθεώρηση, αλλά επιβολή, ε, μεταφορά, μεταφορά του νομοθετικού πλαισίου, παρακολούθηση της επιβολής ε, και, νομοθετη... και συνοδευτικά μέτρα. Επίσης, συμφωνώ και τονίζω αυτά που αναφέρεται για τη δομή. Είχα ζητήσει εγώ το B2B, business to business, να βασιστεί σε μια καθαρή δομή ευρωπαϊκού επίπεδου και πιστεύω ότι αυτό συνάδει και με άλλες οδηγίες σε διαφορετικά επίπεδα και όχι στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Γι' αυτό πιστεύω πριν αναθεωρήσουμε μία οδηγία θα πρέπει να μελετήσουμε ενδελεχώς εάν τα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω της, ε, ε, της ε, λανθασμένης ή της ελλειπούς επιβολής των ομοθετικών διατάξεων. Πιστεύω ότι θίξατε όλα τα σημαντικά θέματα, το ρόλο του Οργανισμού Καταναλωτών, Προστασίας Καταναλωτών, ε, εκεί πιστεύω ότι θα υποβάλω μια τροπολογία ακόμα δική μου. Θέλω να το τονίσω το ρόλο αυτό. Ο Πρόεδρος. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ όλους και τώρα μερικές παρατηρήσεις επειδή είμαι σκιώδης εισηγητής, παρατηρήσεις δικές μου. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχουμε μία συνένεση απόψεων, μία σύμπτωση απόψεων, διότι ήταν ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό μέσο αυτό, το οποίο έτυχε πολιτικής προστασίας ε, τότε, στον καιρό του. Και είναι φιλόδοξο. Είναι φιλόδοξο και σαφώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις στις αγορές. Ακόμα μας απασχολεί το θέμα της συνεπούς επιβολής του νομοθετικού πλαισίου, της εφαρμογής του και της μεταφοράς. Επίσης πρόσεξα ότι το έγγραφο της Κομισιόν τονίζει ορισμένες λίαν ευαίσθητες ε, λίαν ευαίσθητους τομείς πρόσεξα ιδίω ε, το θέμα των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και ξέρω ότι αυτός είναι ένας τομέας που συζητήθηκε σε πρόσφατες διασκέψεις και συνέδρια από πλευράς καταναλωτών και προστασίας καταναλωτών και τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Πιστεύω ότι δεδομένη τη σημασία των περιβαλλοντικών θεμάτων, αύξησης των τιμών κλπ, ε, αυτή όλη η δέσμη είναι πολύ σημαντική. Είναι πιστεύω απογοητευτικό ότι αυτή την πρόταση δεν την πρόσεξαν συνάδελφοί μας από την Περιβαλλοντική Επιτροπή. Έχουμε και τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Αλλά η Επιτροπή Περιβάλλοντος μας στέλνει συνέχεια αμφιλεγόμενες και δύσκολες προτάσεις. Και έχασε την ευκαιρία να σημειώσει εδώ μια καλή δική μας πρόταση. Ε, η άλλη πτυχή που είναι σημαντική είναι η όλη εξέλιξη του συντονισμού της ενημέρωσης και της κυκλοφορίας της ενημέρωσης και την χρησιμότητα της δραστηριότητας SWEEP. Ο, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλα αυτά τα σημεία είχα αναφέρει το θέμα της βαθμολόγησης των ε, καταναλωτών, της βαθμολόγησης από πλευράς καταναλωτών. Ε, την διαχείριση των παραπώνων από πλευράς καταναλωτών, παρακολούθηση ε, των, ε, των προσεγγίσεων, των απόψεων των καταναλωτών, παρακολούθηση της απονομής δικαιοσύνης, δηλαδή της ανταπόκρισης στα δίκαια αισθήματα και αιτήματα των καταναλωτών και την, ε, στο να καταστήσουμε την οδηγία για τις ασέμετες εμπορικές πρακτικές πιο προσβάσιμη στους καταναλωτές, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποφεληθεί από τις διατάξεις που τον ωφελούν ή την ωφελούν. Ε, άλλο ένα σημείο. Συλλογή δεδομένων. Και εδώ η ενημερωμένη και επικυροποιημένη κατάσταση είναι πάντοτε χρήσιμη στη συλλογή δεδομένων. Ε, ως, επίσης την ε, βαθμολόγηση του θέματος από πλευράς καταναλωτών του αν παρακολουθούμε τις, ε, ε, την αθέμητη τιμολόγηση και αν υπάρχουν μεγάλα, ε, μεγάλες διακοιμάνσεις των τιμών. Όταν πήγαμε στην Ελλάδα και σε, μιλήσαμε με προσώπους ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων, μας είπαν ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη ανταγωνισμού διότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και δυνατότητα επέμβασης των καταναλωτών. Ε, ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ροσφόρ για όλα αυτά τα σημεία που έσυξε. Πιστεύω ότι είναι σωστό να διευρύνουμε το πεδίο της πρότασης αυτή και στο B2B business to business και ο τομέας αυτός ε, επιχείρηση προς επιχείρηση ε, θέτει πολλά περισσότερα θέματα, καλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίο από ό,τι απλά των καταναλωτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ε, παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης, το follow-up όπως το κάνουμε πάντοτε, ιδίως όταν μας εφιστά την προσοχή Κομισιόν σε διάφορες απάτες που, που διαπιστώνουμε στην αγορά δεδομένου ότι οφείλονται πολλές φορές σε καταχρηστική ε, διαφήμιση, παραπλανητική διαφήμιση, όπως επίσης και θέματα διασυνοριακά που προκύπτουν. Είναι σημαντικό να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να είμαστε ενημερωμένοι, να παρακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες, ανταλλαγή πληροφοριών και δει στις νέες εξελίξεις, στα περιβαλλοντικά θέματα, στις διαφημίσεις. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα διανύμουμε, να μοιραζόμαστε την πληροφόρηση μεταξύ μας και Επίσης, να ε, χρησιμοποιούμε ό,τι τυχόν μέσον υπάρχει από άλλες δικαιοδοσίες. Οι εμπορικές πρακτικές που ε, διατίθενται στο διαδίκτυο και αυτές μας απασχολούν και αυτές έχουν σχέση άμεση με τις καταναλωτές και γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και το θέμα των παραπώνων ε, που υποβάλλονται στο διαδίκτυο. Πάρα πολλά λοιπόν ενδιαφέροντα θέματα και πιστεύω ότι συμφωνούν και όλοι οι συνάδελφοι ότι στα χέρια του κ. Ροσφόρ το κείμενο αυτό θα βελτιωθεί πολύ με όλες αυτές τις παρατήρησεις. Η κυρία... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ροσφόρ, υπό το φως των καταχρήσεων και των πρακτικών στη χώρα μου, όπως συντοξιούχοι που είχαν ε, επενδύσει σε πρωτισημιακές μετοχές και σε δευτερογενές ε, χρέος και έχασαν όλες ε, τις αποταμιεύσεις τους. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν θεωρείτε ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του 2005 αρκεί προκειμένου τα άτομα αυτά να ε, δουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν επενδύσει γιατί ε, ήταν αντικείμενο, ήταν θύματα ε, απάτης και θέμη των εμπορικών πρακτικών. Γιατί εγώ άκουσα εδώ ότι είπατε να αφαιρεθούν η μαύρη λίστα. Δεν ξέρω αν αρκεί αυτό γιατί τα γεγονότα μας δείχνουν ότι υπήρξαν πολυάριθμες περιπτώσεις και μιλάω για εκατοντάδες οικογένειες που έχουν πληγεί. Δεν μιλώ μόνο για κάποιες σπάνιες περιπτώσεις και καθώς αναλύουμε την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, αυτό που θέλουμε είναι να προβλέψουμε τέτοιες ανεπιθύμητες καταστάσεις και επομένως ε, ρωτώ το γιατί. πρόεδρος αναφέρεστε στην ε, ιδιοκτησία, στα κίνητα ιδιοκτησίας. Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό. Ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Όχι, Πρόεδρε. Αναφέρομαι σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε εμπορικά προϊόντα και σε ε, δευτερογενές χρέος. Um, No. Άλλος κανείς παρακαλώ. Οπότε απευθύνομαι στην Κομισιόν να μας παρουσιάσει τις απόψεις της. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή τη συμπεριστατωμένη, του εμπεριστατωμένου σχεδίου έξεση. Παρουσιάζει ολοκληρωμένα τα θέματα, τα τρέχοντα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμητες πρακτικές. Και η Κομισιόν έχει υποβάλει και τη δική της έκθεση στην αρχή του χρόνου όλοι συμφωνούμε ότι η νομοθεσία αυτή είναι λίαν χρήσιμη, ένα λίαν χρήσιμο μέσο στην εσωτερική αγορά και πολύ ωραίο κιόλα. Και ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα είναι ότι έχει αποδειχθεί κατάλληλο για την αντιμετώπιση προκλήσεων που δημιουργούνται από νέες εμπορικές πρακτικές, κυρίως στον κόσμο του κυβερνοχώρου, του διαδικτύου. Και αυτή είναι η βασική πρόκληση για... που θα έχουμε του χρόνου. Οι αγορές online Έχουμε όλων των ειδών της νέας εξελίξης στο διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, εμπορικές πωλήσει, υπηρεσίες των καταναλωτή, θεμελιώδη δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ούτω καθεξής. παράλληλα με τη σχέδια έκθεση του κυρίου Ροσφόρ, η Κομισιόν έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω προσπάσεις για την ενίσχυση της επιβολής. Και η έκθεση της Κομισιόν τονίζει ότι στο μέλλον θα παίξει ένα ισχυρότερο ρόλο και θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη σε πιο συγκεκριμένους στόχους και θα προσπαθήσει να επιβάλλει έναν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό ε, έλεγχο και επιβολή του νομοθετικού πλαισίου προς όφελος των καταναλωτών. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω όλα τα μέτρα, αλλά θα αναφέρω θα αναφερθώ ειδικά ε, στις, ε, στο σχέδιο έκθεσης και στα σημεία που με απασχολούν. Καταρχάς, το σημείο 4 με 6 του σχέδιου έκθεσης. Η Κομισιόν παρακολουθεί τις ε, εθνικές νομοθεσίες και έχουμε ε, ήδη ένα πλαίσιο επικοδομητικού διαλόγου με τα κράτη-μέλη. Ε, που επίσης εφαρμόζουμε τους δικούς μας έξες, ε, ελέγχους στην ε, μεταφορά της νομοθεσίας όπου δεν καταλήγουμε σε συμφωνία παραπέμπουμε τον παραβάτη στη διαδικασία, στη δικαιοσύνη όπου, όπου σημειώνουμε παρατυπίες και μη συμμόρφωση η Κομισιόν υποστηρίζει μία πιο στενή και στοχευμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν καλύτερα και ταχύτερα σε πολλούς ε, τομείς που αποσχολούν έντονα τους καταναλωτές. Ένα από τα προβλήματα που επηρεάζουν την όλη διαδικασία θέσεις ενισχύει είναι η περιπλοκότητα των διαδικασιών, η έλλειψη συγκεκριμένων κυρώσεων σε παραβάσεις και άλλα. Όμως και ε, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που, που, που σημειώσατε και εσείς όπου η Κομισιόν διαπίστωσε ότι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν παρόμοιες πρακτικές σε διάφορα κράτη-μέλη, όμως ο χειρισμός των δημοσίων αρχών, των κρατικών αρχών είναι διαφορετικός παρόλο που οι περιπτώσεις είναι ίδιες και γι' αυτό υπάρχει το, η, ανείχνευση των πιο ε, συμφερουσών πρακτικών από τους ενδιαφερόμενους από κράτος μέλος σε κράτος μέλος για να δουν που, πρέπει να καταλήξουν για να καταφύγουν στον, στην πιο συμφέρουσα για αυτούς πρακτική. Άρα λοιπόν πρέπει να ε, εδραιώσουμε όλοι μαζί μία ενιαία αντίδραση και ανταπόκριση σε αυτές τις πρακτικές. Στο τέλος Οκτωβρίου στις 29 θα έχουμε σύντομα μια έκθεση για τα ε, ταξίδια και μεταφορές. Επίσης ε, θα έχουμε την αρχή του νέου χρόνου για τις μετακινούμενες ε, κινητές αξίες, ακίνητες αξίες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα σημεία 7 με 9 του σχέδιου έκθεσης που αναφέρει ότι πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο CBC της προστασίας των καταναλωτών. Ε, βάσει του κανονισμού προστασίας καταναλωτών. Ο κανονισμός αυτός, το CPC, δεν προστατεύει μόνο τις διασυνοριακές υπηρεσίες και την διασυνοριακή συνεργασία, που καλύπτουν περίπου το 50% των περιπτώσεων, αλλά ε, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το, να εφαρμοστεί μάλλον αυτό το ε, ο κανονισμός και σε θέματα που αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αναθεώρηση, όπως ξέρετε, του CPC και πιστεύω ότι προς το τέλος του 2014, αρχές του 2015, θα ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση. Έχουμε, κάνουμε ένα δημόσιο, μια δημόσια διαβούλευση προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να να, βρούμε τα, ε, τα νέα κριτήρια, νέες κυρώσεις, ε, ε, διαπίστωση και ταυτοποίηση των παρατυπιών, παραβάσεων, καλύτερη συνεργασία στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών. Όλα αυτά τα σημεία μας απασχολούν στο, στη διαβούλευση. Και τα, η τεκμηρίωση συμβουλευτική τεκμηρίωση μας ε, δείχνει ότι ε, αυτό το έγγραφο ε, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως έγγραφο αναφοράς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από τις αρχές των κρατών μελών. Τώρα λοιπόν η Κομισιόν θέλει να ενημερώσει, να επικαιροποιήσει αυτό το έγγραφο, αυτό το κείμενο. Όπως είπα, πιστεύω ότι θα το έχουμε ολοκληρώσει τον Οκτώβριο του χρόνου. Θα αναφέρει πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Σύγκριση αγορών, τιμών, κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο, δραστηριότητες στο διαδίκτυο, Ε, τιμολόγηση των ταξιδιών και γενικά τιμολόγηση υπηρεσιών στο ταξιδιωτικό τομέα, ε, περιβαλλοντικές πτυχές και ούτω καθεξής. Η Κομισιόν παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ε, διατύπωση και επεξεργασία αυτών των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων. Όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά βασιζόμαστε στην εμπειρία των κρατών μελών για να διαμορφώσουμε την γραμμή μας. Ε, επεξεργαζόμαστε επίσης την, ε, μια τράπεζα δεδομένων η οποία συμβάλλει και αυτή στην καλύτερη επιβολή και συνεργασία και αυτή η τράπεζα δεδομένων αναδιορθώνεται αυτή τη στιγμή και όπως σας είπα την τελευταία φορά τελικά θα καταλήξουμε σε μία διευρυμένη βάση δεδομένων για τον καταναλωτή ε, που θα περιέχει πολύ περισσότερα στοιχεία. Τα στοιχεία τα οποία περιέχει σήμερα δεν περιορίζονται ε, μόνο στην αγγλική γλώσσα, δεν διατυπώνονται μόνο στα αγγλικά, αλλά και σε άλλες ε, γλώσσες θα διατυπώνονται στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως οι βασικές πληροφορίες παρέχονται στα αγγλικά και με τα νέα δεδομένα, δεδομένα θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε και μεγιστοποιήσουμε όλες τις λειτουργικότητες αυτής της βάσης δεδομένων. Ένα σημαντικός τομέας σχετικά με την απόδοση του διεθνού Συστήματος Επιβολής ε, και Εφαρμογής των Κυρώσεων βασίζεται στις ε, παραμέτρους, τους δείκτες επιβολής. Από τη μία πλευρά λοιπόν ε, παρακολουθούμε τις εθνικές νομοθεσίες και από την άλλη παρακολουθούμε την απόδοση εθνικών συστημάτων επιβολής νομοθετικών πλαισίων. Και έχουμε ε, ταυτοποιήσει, έχουμε επισημάνει διάφορους δείκτες ε, με τους οποίους μπορούμε να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε ποιο σύστημα είναι το καλύτερο και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ένα συγκριτικό ε, πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών σε αυτή την ε, κατεύθυνση. Οι κυρώσει είναι σημαντικέ. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στις κυρώσει για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις. Ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη το θέμα αυτό τους απασχολεί και θα παρουσιάσουμε και συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αν μου επιτρέπετε και μου δίνετε χρόνο, Πρόεδρε, θα ήθελα, σας παρακαλώ, να κλείσετε, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, λοιπόν. Ότι σε σχέση με το πρόβλημα business to business, Εργαζόμαστε μια μιας νομοθετικής πρότασης για να απειλήσουμε το θέμα για τους παραπλανητικούς τηλεφωνικούς καταλόγους και ε, θα αναθεωρήσουμε κάποιους κανόνες ε, για να απαγορεύσουν κάποιες πρακτικές και από την άλλη θα συμπεριλάβουμε μέτρα για να ενισχύσουμε το μηχανισμό επιβολής και εφαρμογής νομοθεσίας που έχουν ε, οι επιχειρήσεις για να καταπολεμήσουν αυτές τις απάτες. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ πλήρη παρουσίασή σας, πάρα πολύ νέο υλικό και ιδέες και σίγουρα θα θέλει να τεθετήσει όλα αυτά ο εισήγητης και ίσως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι από αυτών των μέτρων. Γιατί αρχικά η έκθεση, αρχίσαμε τις εργασίες στην έκθεση το Μάρτιο και τώρα θέλουμε να προσπαθήσουμε να δούμε αν έχουν υπάρξει και νέες εξελίξεις από τότε. Ο κύριος Ροσφόρ, παρακαλώ. Θέλετε να συνοψίσετε για τα όσα υπόθηκαν, τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα και να μας πείτε και ποιο είναι και το χρονοδιάγραμμα για το επόμενο στάδιο των εργασιών σας. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτη παρατήρηση. Σας ευχαριστώ φυσικά για τις συνεισφορές σας και διαπιστώνω ότι είναι συγκλίνουσε όλοι οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση και επομένως από τη σκοπιά αυτή θα είναι εύκολο να βελτιώσω το κείμενο με τροπολογίες που θα λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις. Γενικά πιστεύω ότι είμαστε σύμφωνοι. Θα ήθελα να, να απευθυνθώ στον κύριο Μπόρισεφ. Έχει δίκιο να επιμένει για την πρόληψη, αλλά τελικά όταν επιμένει σε αυτό, αιτιολογεί ότι πρόκειται για μια οδηγία μέγιστη εναρμόνισης. Και εδώ αναφέρομαι και σε αυτό που τόνισαν πολλοί συνάδελφοι και η κυρία Σενάλοβα ανεφερθήκε στην διασυνοριακή λογική. Η μέγιστη εναρμόνιση επιτρέπει να κυκλοφορούν πολύ καλύτερα οι πληροφορίες. Δηλαδή, έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε διαφήμιση γύρω από τις πρακτικές που δεν είναι πλέον δυνατές και υπάρχουν σε αυτό το κατάλογο που είναι ο ίδιος για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το σημείο επιμένω. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε την πρόληψη αυτή, αλλά στο καθιστά δυνατό αυτό η μέγιστη ενερμόνιση. Όμως φυσικά δεν θα πρέπει να μεταφραστεί σε απώλεια προστασίας για τους καταναλωτές. Η κυρία Πέρες αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει από τον τύπο, δηλαδή για το τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι που ζουν ε, εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σήμερα. Νομίζω ότι αυτή η οδηγία δεν ε, θίγει ε, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες στον τομέα των κινήτων, ε, γιατί ουσιαστικά εμπίπτουν σε μια άλλη σφαίρα. Πέρα από την καθαρή κατανάλωση αφορούν την απόκτηση κεφαλαίου. Κυρία Πέρες, η κυρία Πέρες αναφέρθηκε σε μία μείωση του περιεχομένου του μαύρου καταλόγου, της μαύρης λίστας. Όχι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Πρέπει απλώς να διασφαλίσουμε και η Κομισιόν άλλωστε όταν αναφέρθηκε στις προσπαθίες της για τη βελτίωση του εγγράφου προσανατολισμού δεν μας καθησύχασε ακριβώς, αλλά μας παρουσίασε κάτι που συνάδει με αυτό που θέλουμε, δηλαδή την αναθεώρηση αυτού του εγγράφου προσανατολισμού, έτσι ώστε τελικά να υπάρχουν πολύ λιγότερες αποκλίνουσες ερμηνείες επί αθέμητων πρακτικών ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Και κάτι που με εκπλήσει ιδιαίτερα ακούγοντα τις διάφορες παρατηρήσεις είναι ότι τελικά βλέπουμε πως σιγά σιγά οικοδομούμε ένα συνεκτικό οικοδόμημα όταν Πρόκειται, και εδώ το ανέφερε η κυρία Σενάλοβα αυτό, όταν πρόκειται ε, για τα διασυνορικά ζητήματα, όταν επιμένουμε ιδιαίτερα σε αυτά και για τις επιγραμμικές πωλήσει, επισέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία όταν είπατε ότι μπορεί παραδείγματο χάρη να μην ξέρουμε που βρίσκονται διάφοροι εμπορευόμενοι και να μην έχουμε τα στοιχεία τους. Εδώ δεν ε, απαντάμε ε, στην οδηγία των δικαιωμάτων καταναλωτών στα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να έχουμε ένα συνεκτικό οικοδόμα και το ίδιο ισχύει για το ADR και το ODR. Αυτή η διαδικασία επίσης συνεχίζεται Ουσιαστικά ε, αντιμετωπίζοντας ε, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ε, εδώ η Κομισιόν θα οργανώσει κάποια σεμινάρια για να διαδώσει τις βελτιστές πρακτικές. Ο κύριος Χάρμπορ έχει δίκιο που επιβαίνει στα περιβαλλοντικά θέματα και Σήμερα έχουμε ουσιαστικά ε, ένα τρόπο να ε, διαδοθεί ε, αλλά με λανθασμένο τρόπο αυτό το περιβαλλοντικό επιχείρημα και να οδηγηθούμε σε αθεμίτες πρακτικές. Τώρα για το B2B αναφέρθηκε σε αυτό και η κυρία Ρούλα και ο κύριος Χάρμπορ και η Κομισιόν. Είναι σαφές ότι για μας θα πρέπει το business to business να το αφορά αυτή η καταγγελία τώρα θέμα των πρακτικών, όμω, το θέμα είναι σε ποιο νομοθετικό όχημα θα γίνει αυτό. Η οδηγία που συζητάμε σήμερα, και το επενθύμησαν πολύ, ο κύριος Μπόρισοφ έτσι ξεκίνησε την παρέμβασή του, εφαρμόζεται με τόσο κατακαιρματισμένο τρόπο που μου φαίνεται δύσκολο ε, να επεκτείνουμε αμέσως το πεδίο εφαρμογή με τον B2B. Ας μην ξεχνάμε ότι στην οδηγία αυτή ε, υπάρχει διορισμένη μία αρμόδια οντότητα σε κάθε κράτος μέλος για την εφαρμογή της οδηγίας και αυτή η οντότητα ταυτόχρονα μπορεί να ασχολείται και με το B2B και με το B2C και τότε έχουμε δυσκολίες γιατί δεν μιλάμε για τις ίδιες διοικητικές υπηρεσίες ούτε για τις ίδιες τους οργανισμούς. Και επιμένουμε, το πενθύμησαν και στους στήλιστες συνάδελφοι, για την ανάγκη να υποστηρίξουμε την προστασία των καταναλωτών, όμως πολύ συχνά έχουμε διαφορετικά όργανα που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών ε, και άλλα που ασχολούνται με το B2B. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει και B2B να ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, αλλά σίγουρα αυτό δεν θα γίνει στο ενδεχόμενο πλαίσιο αυτής, της αναθεώρησης αυτής της οδηγίας και θα πρέπει μία μέρα να δούμε και το C2C που αναπτύσσεται πολύ σήμερα ε, με το ίντερνετ, δηλαδή από καταναλωτή σε καταναλωτή. Πολλέ ε, φορέ ε, και οι καταναλωτέ γίνονται πολιτέ, αλλά όλα αυτά δεν είναι ρυθμισμένα από την νομοθεσία, είναι ένα άγνωστο πεδίο που θα πρέπει να το προσεγγίσουμε, γιατί όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε καταναλωτέ που πολλούν προϊόντα και μπορεί να είναι και εκεί να συναντάμε θέμητε πρακτικές. Περιμένω λοιπόν με πολύ ανυπομονησία και ενδιαφέρον τις τροπολογίες ε, που θα μου στείλετε. Η προθεσμία είναι πολύ σύντομη γιατί έχει καθοριστεί στις 23 Οκτωβρίου. Θα τις εξετάσουμε τη συνεδρίαση μας 27 ε, και 28 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία προβλέπεται στην Επιτροπή 12, ε, συγγνώμη, 17 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Yes, well, thank you very much indeed. Um... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε προθεσμία μέχρι τις 23 για τις τροπολογίες όπως είπατε και έχουμε χρόνο για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που ήρθε για το θέμα αυτό. Προχωρούμε λοιπόν μία πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή στη ζωή της Επιτροπής μας είναι η τωρινή, γιατί θα ξεκινήσουμε την εξέταση μιας νέας πρότασης, την οποία περιμέναμε όλοι εδώ και πολύ καιρό. Ε, ο πύχης των προσδοκιών είναι ψηλά και χαίρομαι διότι μπορώ επισήμως να καλωσορίσω την κυρία Μανφρέιντι, επικεφαλής ε, του τμήματος και τον κύριο Κώστα Πέτρου, πολύ γνωστό, ενεργό συμμετέχοντα της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, που έχει πάρει το λόγο για πολλούς και διαφορετικούς φακέλους εδώ και πολλά χρόνια, θα μας παρουσιάσει την αξιολόγηση αντικτύπου και θα συζητήσουμε την έναρξη της διαδικασίας. Καλωσορίζω και τον Hans Peter Mayer, τον ε, προσφάτως ε, διοριστέντα εισηγητή μας. Πρώτη φορά θα παίξει αυτό το ρόλο σήμερα το απόγευμα. Έχουμε απουσία σκιωδών εισηγητών σήμερα, εκτός από την κυρία Μακλάρκιν Εγώ θα τα παρακολουθήσω αυτά και η κυρία Ρούιλε. Ε, θα κρατήσουμε σημειώσεις και θα τα διαβιβάσουμε στους ε, σκιώδεις εισηγητές και ο κύριος Γοσφόχ ενδεχομένως για τους φιλελεύθερους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θέσουμε ερωτήματα για την πρόταση αυτή. Ποιος θα παρουσιάσει ο κύριος Πέτρου? Νομίζω ότι έχετε φέρει διαφάνειες, θα πρέπει να τις ετοιμάσει ο τεχνικός για να τις προβάλλει και με χαρά θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ διότι δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρόταση ε, οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και την αξιολόγηση αντικτύπου που προηγήθηκε της πρότασης. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κύριο Hans Peter Μάιερ για τον ε, διορισμό του ως εισηγητή σε αυτό τον πολύ σημαντικό φάκελο. Σωστά λέτε κύριε Πρόεδρε, ήταν μια πρόταση την οποία περιμέναμε όλοι εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε ολοκληρώσει μια αρκετά εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης και όταν την ολοκληρώσαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή νιώσαμε έτοιμοι να υποβάλουμε μία πρόταση. Η διαδικασία η διαβούλευση είχε ξεκινήσει το 2007, συνεχίστηκε το 2008. Αυτά τα έτη έλαβε χώρα η πρώτη διαβούλευση. Στη συνέχεια η Κομισιόν εκπώνησε μία μελέτη ε, για τα οργανωμένα ταξίδια, ε, για το αν αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή, για τα νέα προϊόντα που έχουν ε, εισαχθεί στην αγορά. Στη συνέχεια είχαμε ένα δεύτερο γύρο διαβούλευσης το 2009 με πάρα πολλά εργαστήρια, πάρα πολλά συνέδρια ε, όπου θελήσαμε να πάρουμε τη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων, των κρατών μελών, των επισήμων αρχών. Το 2012 έγινε η αξιολόγηση αντικτύπου και το 2013 επιτέλους τον Ιούλιο παρουσιάστηκε η πρόταση, όπως τα γνωρίζετε όλοι. Επομένως, τι θέλουμε να πετύχουμε με την πρόταση αυτή για μια νέα οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα σας πω αμέσως. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει και το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο σε, για κανέναν από εσά. Η αγορά των ταξιδίων έχει εξελιχθεί πολύ από τότε που υιοθετήθηκε η φυστάμενη οδηγία στη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Και αυτό κυρίως οφείλεται στην επανάσταση του διαδικτύου, στην ηλεκτρονική επανάσταση, στη δυνατότητα που έχουν οι ταξιδιώτες και οι καταναλωτές να κλείνουν μόνοι τους τα εισιτήριά τους και να οργανώνουν μόνοι τους τα ταξίδια τους στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι που τάραξε σε βάθος τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά και άλλαξε άρδιν την κατάσταση. Μείωσε σημαντικά τον αριθμό των πακέτων, ε, των ταξιδιωτικών πακέτων που είχαν οργανωθεί εκ των προτέρων, που ήταν και κυρίαρχα στον κλάδο, στην αγορά την τουριστική, πριν ε, τεθεί σε ισχύ η οδηγία αυτή. Η κατάσταση σήμερα πώς έχει. όλη η αγορά διακοπών καταμερίζεται όσο εξής. Το 54% των καταναλωτών κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις και διευθετήσεις, κλείνουν δηλαδή μόνοι τους όλα τα κομμάτια του ταξιδιού τους. 23% μόνο αγοράζουν τα παραδοσιακά τουριστικά ταξιδιωτικά πακέτα που προσφέρουν οι tour operator και που πολλούνται μέσα σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο ή μέσα από ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Και το υπόλοιπο 25-26% περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε αυτό το ποσοστό ο καταναλωτής συνθέτει από μόνος του, φτιάχνει έναν συνδυασμό διαδικτυακά για το ταξίδι του. Ε, είναι συνδυασμένες ε, ρυθμίσεις ταξιδιωτικά, τις αξιδιωτικές με έναν έμπορο. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής επισκέφτεται ένα site που προσφέρει τη δυνατότητα να κλείσει και το ταξίδι και τη στέγαση μαζί. Κλείνει λοιπόν το ταξίδι, τα εισιτήρια κτλ. Ή μάλλον ε, διορθώνω λέει ο μιλήτης, επιλέγει π.χ. μία πτήση και ενδεχομένως επιλέγει, επιλέγει και τη στέγαση στον ε, τόπο προορισμού και κάνει check-out μετά και πληρώνει και για τα δύο αυτά σκέλη των διακοπών του με τη μία. Είναι μια κατάσταση ας πούμε ε, καλαθιού αγορών. Η Expedia είναι ένας operator, ένας φορέας που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Όμως Έχουμε και άλλες καταστάσεις όπου κανείς μπορεί, για παράδειγμα, να κλείσει ένα ταξίδι, μια πτήση και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής του ζητείτε ή ενθαρρύνεται αυτός που κλείνει την πτήση να προσθέσει και ενοικίαση αυτοκινήτου ή ε, κλείσιμο δωματίου σε ξενοδοχείο από κάποιον άλλον έμπορο, από κάποιο άλλο website, αλλά υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο site και ο καταναλωτής αν τελικά το εγκρίνει και αποφασίσει να τα επιλέξει όλα, πληρώνει με τη μία το σύνολο του ποσού που επιμερίζεται στα site που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Βέβαια οι περιορισμοί εδώ είναι πολύ πιο χαλαροί για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να μην πληρώσει με τιμία το τελικό σύνολο, αλλά καλείται να διευθετήσει και να ρυθμίσει το δεύτερο τμήμα της κράτησης ε, αφού πλοηγηθεί σε ένα άλλο ανεξάρτητο site. Υποβοηθούμενες δηλαδή ταξιδιωτικές διευθετήσεις, πρόγραμμα ε, τουρισμού που στηρίζουν και υποβοηθούν διάφορα ε, site και διάφοροι έμποροι, εταιρείες που εμπορεύονται αυτά τα πράγματα. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση καλύπτει το 26% της αγοράς, 17% είναι το πακέτο το διαδικτυακό με έναν έμπορο, με ένα site που πουλάει και την, ε, το ταξίδι και τη στέγαση και όλα. Επομένως, Ε, πρόκειται για εξελίξεις πολύ σημαντικές. Τις παρατηρήσαμε, αναλύσαμε την αγορά, διαβουλευθήκαμε με τους εμπλεκόμενους φορείς και με τα κράτη-μέλη. Σημειώσαμε λοιπόν και παρατηρήσαμε το εξής. Η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια δεν καλύπτει αυτές τις νέες υπηρεσίες και μάλιστα δημιουργεί και προβλήματα στην αγορά. Ε, δημιουργεί και προβλήματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές. Τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις απαριθμώνται λεπτομερώς στην αξιολόγηση αντικτύπου που κάνουμε και είναι τριπλής διάστασης, τριών διαστάσεων. Δεν είναι παιχνίδι επί ίσης όρης. Οι συνδυασμένες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο διαδίκτυο φαίνονται σαν οργανωμένα ταξίδια πακέτο ε, στον καταναλωτή, αλλά δεν συμμορφούνται και με αυτούς τους κανόνες. Και άρα υπάρχει θέμα με το κόστος συμμόρφωσης το οποίο δεν υποχρεωμένοι οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών να αναλάβουν, ενώ το κάνουν τα, τα παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία με τα πακέτα που προσφέρουν. Και είναι ένα κόστος που, έχει να κάνει με τα, που φτάνει μέχρι 10 ή 12 ευρώ ανά πακέτο. Άρα άνηση, ε, άνισος, ε, άνιση όρη για δύο κλάδους οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε και είδαμε ότι η 12 ευρω ανα πακετο αρα ανηση ανισος ορη για δυο κλαδους οι οποιοι ανταγωνιζονται μεταξυ τους απο εκει και περα πιστευουμε και ειδαμε οτι η οδηγια του 1990 περιλαμβάνει προαπαιτούμενα τα οποία είναι παροχημένα και συνεπάγονται κόστος συμμόρφωσης ε, υψηλό ή μη δικαιολογημένο. Για παράδειγμα, ε, προϋποθέσεις ενημέρωσης που έχουν να κάνουν με τα φυλάδια και αυτές οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ δαπανηρές για τις ε, επιχειρήσεις. Στην εποχή του διαδικτύου δεν φαίνονται να είναι απαραίτητες οι ρυθμίσεις αυτές και αν υπάρξει ένα streamlining όλων αυτών, μια ευθυγράμμιση, μια συμμόρφωση, θα επιτευχθούν και οι οικονομίες. Η σημερινή οδηγία, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή, προστατεύει τους ε, όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και δεν εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο στα κράτη-μέλη. Όμως στο πεδίο εφαρμογής της αναφέρεται ότι έτσι εφαρμόζεται και δεν ισχύει αυτό στην πράξη, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Και συνεπάγεται κόστος συμμόρφωσης ε, για περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται προστασία. Όταν, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις κλείνουν ε, τα ταξίδια τους μέσω μιας εταιρείας διαχείρισης ταξιδίων και έχουν συνάψει με αυτή την εταιρεία συμφωνίες πλαίσιο. Και τρίτον, το γεγονός ότι η οδηγία αυτή βασίζεται στην ελάχιστη εναρμόνιση είναι κάτι που οδήγησε σε πολλούς και διαφορετικούς αποκλίνοντες κανόνες μεταξύ των κρατών μελών και όσοι, όσες εταιρείες και φορείς θέλουν να λειτουργήσουν διασυνοριακά πρέπει να ευομιστούν επιπρόσθετα βάρη, επιπρόσθετο κόστος για να συμμερφωθούν με, τις, με τα απαιτούμενα, τα προαπαιτούμενα σε κάθε κράτος μέλος. Από εκεί και πέρα. Στην αξιολόγηση αντικτύπου σε όλη αυτή τη διαδικασία αξιολογήσαμε το βάρος για τον καταναλωτή των παραδοσιακών οργανωμένων ταξιδίων σε σύγκριση με τις νέες αυτές δυνατότητες. Μιλούμε ε, δηλαδή για τα μη προστατευμένα τουριστικά ή ταξιδιωτικά αγαθά και το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο, 593 ευρώ σε σχέση με 100 τόσα ευρώ ε, ε, την, την, την άλλη πλευρά. Επομένως, το βάρος για το καταναλωτή μπορεί να είναι μεγαλύτερο, πιο δαπανηρό. Οι κανόνες δεν είναι παρκείς, δεν είναι αρκετά καλοί, δεν διασφαλίζουν σωστή προστασία του καταναλωτή. Μπορεί να είναι και απειρχαιωμένοι και παροχημένη, κάτι το οποίο ε, είναι σε βάρος του καναλωτή επίσης. Και εδώ αναφέρομαι στην οδηγία που επιτρέπει αύξηση τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν λέει πόσο, μέχρι πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές. Η, η αβεβαιότητα οδηγεί σε έλλειψη σαφήνειας για τον καταναλωτή και ως προς την αποζημίωση η ηθική βλάβη ε, δεν εξηγείται σαφέστατα από την πρόταση και αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ πολλών. Επομένως, από τη στιγμή που υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, αποφασίσαμε να καθορίσουμε στόχους πολιτικής για την πρόταση αυτή. Και πρώτος γενικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον ε, ταξιδιωτικό κλάδο οργανωμένων πακέτων ταξιδίων. Και εδώ υπάρχουν τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε ε, περισσότερο ισότιμες συνθήκες για τις επιχειρήσεις, να ενθαρρύνουμε διασυνοριακές προσφορές και να μην υπάρχει ε, κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις το οποίο να μην δικαιολογείται, να πρέπει να το επομιστούν και μάλιστα αδίκως. Θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά και οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι. Να μειώσουμε το βάρος που επομίζεται ο καταναλωτής έχοντας περισσότερη διαφάνεια και προσφέροντας περισσότερη προστασία σε αυτά τα νέα ε, ταξιδιωτικά αγαθά, τα συνδυασμένα. Και θέλουμε να πλουστεύσουμε τους υφιστάμενους κανόνες, να είναι πιο εύκολο για τον καναλωτή να επιζητήσει βοήθεια ή και αποκατάσταση ε, του προβλήματος και της βλάβης που του έχει προκληθεί. Η αρχή της αναλογικότητας ισχύει πάντοτε, όπως γνωρίζετε, και παρά τις αποκλήσεις μεταξύ εθνικής νομοθεσίας των διαφόρων κρατών μελών, δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να είναι αντικειμενικά, θα παραμείνουν τα εμπόδια. Δηλαδή, εάν αφήσουμε τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με αυτό το θέμα μόνα τους, εκτός ευρωπαϊκής αρμοδιότητας δηλαδή, θα καταλήξουμε σε ακόμα μεγαλύτερο κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς. Έχουμε λοιπόν οκτώ επιλογές πολιτικής. Η πρώτη είναι να παραμείνει το status quo. Δεύτερη, να εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα εφαρμόζεται η οδηγία σε νέες καταστάσεις και να βελτιώσουμε την εφαρμογή της. Τρίτη επιλογή, να θεσπίσουμε συγκεκριμένη σήμανση και ετικετοθυσία των οργανωμένων ταξιδίων και των πακέτων για την ενημέρωση του καταναλωτή. Τέταρτον, να ανακαλέσουμε την οδηγία και να την αντικαταστήσουμε με κανονισμό. Πέμπτη επιλογή νομοθετική επιλογή. Να εξυγχρονίσουμε την οδηγία, να τη διευκρινίσουμε και να διευρύνουμε το πεδίο που καλύπτει για να περιλάβει και τα οργανωμένα ταξίδια από μία επιχείρηση τα οποία τα προτείνει ως υπηρεσία διαδικτυακά. Έκτη επιλογή, διαβαθμισμένη προσέγγιση σταδιακή, δηλαδή περιλαμβάνει το 5, να περιλάβουμε δηλαδή και τα πακέτα, τα οργανωμένα ταξίδια από μία εταιρεία, αλλά και την υπηρεσία την ταξιδιωτική και τα ταξιδιωτικά προϊόντα που προσφέρονται από διαφορετικές ε, διαδικτυακές εταιρείες, υποβοηθούμενες ε, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις που υπάγονται σε ένα πιο ελαφρό, ε, λιγότερο άκαμπτο νομοθετικό πλαίσιο. Έβδομη επιλογή είναι πλήρη κάλυψη όλων αυτών των πακέτων και των οργανωμένων ταξιδίων και ρυθμίσεων. Μία μαξιμαλιστική δηλαδή προσέγγιση. Και η όγδοη επιλογή είναι μία οδηγία για όλα τα ταξίδια που να καλύπτει όλες τις ταξιδιωτικές ή τουριστικές υπηρεσίες. Την απορρίψαμε την 8η επιλογή στην αξιολόγηση αντικτύπου για τους εξής λόγους. Οι ανεξάρτητες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, το γεγονός δηλαδή ότι ο καταναλωτής κανονίζει μόνος του, γιατί στο 8 θα έπρεπε να, να μπουν ε, και αυτά στην οδηγία, δηλαδή όταν κάποιος κλείνει ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο μόνος του, ως καταναλωτής. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι εκτεταμένη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία καλύπτει ε, τους ανθρώπους που, κάνουν, που κανονίζουν μόνοι τους. Έχουμε την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές, έχουμε την οδηγία για τους καταναλωτές που θα αρχίσει να ισχύει ΛΙΑΝ σύντομα και έχουμε και διάφορους κανονισμούς στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών. Καλύπτονται λοιπόν όσοι κάνουν το ε, δικό τους πρόγραμμα ατομικά, ανεξάρτητα. Ο καταναλωτής γνωρίζει ξεκάθαρα με ποιον έχει να κάνει, ποιος είναι ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών, άρα δεν δυσκολεύεται τόσο ενώ όταν μιλούμε για οργανωμένα ταξίδια ή πακέτα, ένας άνθρωπος είναι που συναρμολογεί αυτό το πακέτο και του το προτείνει στον καταναλωτή, αλλά είναι πιο σκοτεινό πώς, ποιος ακριβώς κρύβεται από πίσω και πώς είναι αυτή που υπάρχει αυτών των υπηρεσιών και είναι δυσκολότερο να κάνει αξιολόγηση. Απορρίψαμε λοιπόν την 8η επιλογή και μας έμειναν οι πρώτες 7. Εξετάσαμε την πρώτη επιλογή, να διατηρηθεί το status quo και να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση, το βαθμό συμμόρφωσης με τις οδηγίες, ποιο είναι το κόστος ε, των ε, διασυνοριακών εμπορικών δραστηριοτήτων 1,65 ευρώ ανά πακέτο οργανωμένο ταξίδι αυτό είναι το κόστος για τη διασυνοριακή προσφορά αυτής της υπηρεσίας θεωρήσαμε λοιπόν ότι τεκμηριώνεται η ανάγκη να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την κατάσταση και να προσφύγουμε στις άλλες επιλογές, από 2 ως 7. Η δεύτερη που έχει να κάνει με τις κατευθυντήριες γραμμές. Την αξιολογήσαμε αυτή την επιλογή και συμπεράναμε ότι δεν θα μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις και να το κάνουμε. Τα προβλήματα θα παραμείνουν και πολύ λίγοι εμπλεκόμενοι φορείς σε όλες τις διαβουλεύσεις τη στήριξαν ως επιλογή. Τώρα, ως προς την τρίτη επιλογή που είναι η σήμανση των προϊόντων αυτών, η ετικετοθεσία αν θέλετε, θα αυξηθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις με σχετικά μικρό αντίκτυπο στον καταναλωτή ευεργετικό. Η μελέτη μας έδειξε ότι μόνο το 3% των καταναλωτών θα κάνουν κλικ σε αυτή την σήμανση η οποία θα περιλαμβάνει τα δικαιώματά τους. Ανάκληση της οδηγίας, τέταρτη επιλογή οδηγεί σε, πολλές, σε μεγάλη εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις, προφανώς 10 ή 12 ευρώ ανά πακέτο που προσφέρεται εξοικονομείται από την επιχείρηση, όπως ήδη σας είπα. Ωστόσο θα αυξηθεί πολύ το κόστος που αναλαμβάνει ο καταναλωτής γιατί θα καταργηθεί το καθεστώς προστασίας του καταναλωτή. Η μια απορρίθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ενισχύσει το νομικό κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά. Ε, τα κράτη-μέλη ε, θα ε, προβλέψουν κανόνες ελεύθερα ο καθένας, το κάθε κράτος μέλος τον δικό του, χωρίς να υπάρχει ομοιογένεια. Τώρα, ως προς την πέμπτη επιλογή να ε, καλύψουμε μόνο τα οργανωμένα ταξίδια που προτείνονται από έναν trader, να διαγράψουμε και να αφαιρέσουμε τους κανόνες για τα φυλάδια. Αυτό είναι καλό. Θα μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις κατά λίγα ευρώ, το οποίο τελικά ε, θα αθρίσει, θα κάνει να αθρηστεί ένα μεγάλο ποσό, θα αυξηθεί το κόστος συμμόρφωσης αφού και νέα προϊόντα θα μπουν κάτω από το πέπλο της νομικής αυτής κάλυψης και προστασίας, τελικά θα έχουμε εξοικονόμηση συνολικά 80 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την έκτη επιλογή που εξετάσαμε, περιλαμβάνει την 5 που έχει μόνο τον έναν trader, αλλά και τις υποβοηθούμενες ταξιδιωτικές διευθετήσεις και ε, τα οργανωμένα ταξίδια από πολλούς trader. Θα γίνουν οι ίδιες εξοικονομήσεις όπως στην επιλογή 5, αλλά θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο ανταγωνισμός, γιατί πολλά περισσότερα τουριστικά προϊόντα θα μπουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αλλά θα υπάρξει και βελτιωμένη ευελιξία σε σχέση με την πέμπτη επιλογή, διότι επιχειρήσεις είτε που πολλούν με, έναν trader ή με πολλούς trader, ε, με έναν trader για παράδειγμα η Expedia μπορούν εύκολα να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να πάνε προς το ε, να προσφέρουν υποβοηθούμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και άρα να απολαύσουν ενός πιο ελαφρού νομοθετικού πλαισίου και αντιστρόφως. Θεωρούμε ότι το 25% των ε, οργανωμένων ταξιδίων με έναν trader και το 35% των ε, οργανωμένων ταξιδίων με πολλούς τρέιντερ θα ε, προσαρμοστούν υπ' αυτή την έννοια. Και αυτό θα μειώσει το επιπρόσθετο κόστος συμμόρφωσης γιατί προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή υπαριθμών 6 είναι προτιμητέα, είναι αυτή που προτιμούμε και γι' αυτό η πρόταση που υποβάλλουμε βασίζεται στην έκτη επιλογή που εξετάσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πλήρη επισκόπηση και Μπορώ να σας πω, μας δείχνει τι πρέπει να κάνει μια ποιοτική μελέτη εκτίμηση επιπτώσεων να αναλύσει όλες τις επιλογές και κάνατε μια πλήρη δουλειά στην περίπτωση αυτή και πραγματικά μπόρεσα να παρακολουθήσω την προσέγγιση των οκτώ επιλογών. Όμω εγώ νομίζω ότι η παριθμόν 6 επιλογή φαίνεται να επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία και φαίνεται να έχει γίνει αποδεκτή κυρίως σε χώρες όπως είναι η δική μου. Και ξέρετε πάρα πολύ ε, ταξιδιώτες που αγοράζουν αυτά τα πακέτα προέρχονται από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή ίσως ε, για να θέσει κάποιες ερωτήσεις αν το επιθυμεί και κατόπιν ε, θα σας παρακαλούσα να παρουσιάσετε και το χρονοδιάγραμμα, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Να καλωσορίσω και τα νέα μέλη. Παρακαλώ, ο εισηγητής έχει το λόγο. Και το ε, αυτής της πλήρους παρουσίασης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κομισιόν για αυτή την ε, εμπεριστατωμένη παρουσίαση της ε, μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων. Τα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να δω πώς θα τα πάμε με την έκτη επιλογή, την έκτη οψιόν η οποία παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις ή εάν μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και ορισμένα στοιχεία από τις άλλες οψιών. Όταν παρουσίασε την 1η Ιουλίου η Κομισιόν, οι συντονιστές τότε και σήμερα, ε, τότε αποφάσισαν ε, την ανάθεση ε, του, της έκθεσης και βλέπετε σήμερα ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και μέχρι το Μάρτιο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία αυτού του θέματος για να μπορέσει να ψηφιστεί στην πρώτη Ολομέλεια. Ε, η Ολομέλεια του Ιουλίου ε, θα είναι βεβαρημένη με τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα τα οποία υπήρχαν πριν από τις εκλογές. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε μόνο εάν συνεργαστούμε σωστά, εάν οργανωθούμε και συντονιστούμε από κοινού και η γραμματεία έχει προχωρήσει περισσότερο, είναι πιο προχωρημένη επειδή ασχολείται με το θέμα από καιρό. Χαίρομαι για τη συνεργασία μαζί τους και χαίρομαι και για τη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές διότι παρόλες τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί έναντί μου, εμού, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ ε, σωστό λογικό συμπέρασμα και έτσι μετά από την ακρόση της 5ης Νοεμβρίου θα ήθελα να οργανώσω ένα, μια πρώτη συνάντηση των εισηγητών ώστε να μπορέσουμε έγκαιρα να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε. Τώρα, τι πιστεύουμε εμείς, ποια είναι η δική μας άποψη. Είναι οι ορισμοί, είναι το πεδίο εφαρμογής, είναι τα δικαιώματα και οι απαιτήσει των ε, ταξιδιωτών, είναι οι οι ευθύνες, είναι οι διαδικασίες αναχώρησης και άφηξης και είναι και εθνικές διατάξεις. Πιστεύω ότι η απορρίσμηση της ε, αεροπλοείας των αεροπορικών μεταφορών έχει αυξηθεί σημαντικότατα μετά από τον τελευταίο κανονισμό και επίσης είναι δεδομένο ότι έχουν αλλάξει εντελώς οι τρόποι ε, με τους οποίους οργανώνουν οι ταξιδιώτες τις διακοπές τους. Γι' αυτό με την Κομισιόν συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχουν ακόμα διάφορες ασαφείς, διάφορες γκρίζες ζώνες οι οποίες δεν ξέρουμε αν εμπίπτουν την οδηγία ή όχι και γι' αυτό χρειάζεται, ε, χρειάζονται πολλές ευκρινήσεις και σαφήνεια και διαφάνεια. Υπάρχει μία νομική βάση η οποία είναι ανομιογενής, δεν είναι ενιαία. Πρέπει να την προσαρμόσουμε λοιπόν. Ε, επίσης υπάρχει το θέμα των επιχειρήσεων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά και ε, δυστυχώς υποβάλλονται σε περιτά έξοδα τα οποία δεν είναι αναγκαία. Πέραν αυτού έχουμε και μία υποχρέωση ενημέρωσης, ε, ε, αλλαγή των, ε, του νομοθετικού πλαισίου πριν από την αναχώρηση, ειδικά έναν πλήρη έλεγχο το, της διαδικασίας αποζημιώσεων σε περίπτωση που χρεοκοπεί ένα ταξιδιωτικό γραφείο και τη διαδικασίας στήρισης των αμοιβαίων υποχρεώσεων και των δύο πλευρών. Επίσης, ήδη μπορώ να ανακοινώσω ότι ιδιαίτερα ο σεβασμός των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τις συμβάσεις, τις υποχρεωτικές συμβάσεις, θα αποτελέσουν ένα κεντρικό σημείο της έξεσης μου. Διότι, ξέρετε ότι όσον αφορά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών τώρα, είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος και συγχαίω, ε, ε, συγχίζομαι Κάθε φορά που μια αεροπορική εταιρεία λέει ότι άμα δεν μου, πάνε, δεν μου ταιριάζουν οι συνθήκες ή δεν έχω αρκετούς επιβάτες ή δεν μου γουστάρει να <laughs> κινήσω το αεροπλάνο, ακυρώνω την πτήση αυτό με θυμώνει ιδιαίτερα, διότι τα επιχειρήματά τους ε, όχι μόνο δεν είναι βάσιμα, αλλά είναι απαράδεκτα. Ε, όποτε θέλουν λοιπόν παραβιάζουν την συμβατική, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και απειλούν ε, όχι μόνο τους ταξιδιώτες αλλά και τα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ε, αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, παρατυπίες και θα είμαι πολύ σκληρός ε, εναντί τους, αλλά θα είμαι και πάρα πολύ σωστός εναντί των εταιριών που συμπεριφέρονται σωστά. Τώρα το χρονοδιάγραμμα έχει λίγο αλλάξει από το αρχικό. Δεν θα πω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά στις 5 δεκάτου, δεδομένου ότι έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα ακρόση, θα έχουμε τη δυνατότητα μια εμπειρία ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Good. Um... Πρόεδρος. Κύριε Ρου... Ρούλε, όχι, Ρούλε, όχι, δεν θέλω να παρέμβω. Ο πρόεδρος, να σχολιάσω κι εγώ και μερικές ερωτήσεις στην Κομισιόν. Πιστεύω ότι έχετε βρει τη σωστή ισορροπία, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ πολύ διάστατη η φύση των ταξιδιών και των ταξιδιωτικών μετακινήσεων. Ε, μιλάμε πολύ για τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροπορικά ταξίδια. Και μην ξεχνάτε ότι συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών που και τους απασχολούν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, του επαναπατρισμού, στις αλκοολικές ε, μεταφορές και έχουν <laughs> σημαντικά αλλάξει τις απόψεις τους από τότε που ξεκίνησε η αρχική διαδικασία με την πρόταση. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες πτυχές της αρχικής ταξιδιωτικής ε, οδηγίας τα οποία καλύπτονται αυτή τη στιγμή αλλά αναρωτιέμαι εάν ορισμένα συγκεκριμένα σημεία πρέπει να θεωρηθούν έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή και συνέπεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι από την αρχική οδηγία ταξιδιωτικών ομαδικών ταξιδιών, πακέτων, έχουμε δει να διευρύνεται σημαντικά η κίνηση στους αυτοκινητόδρομους υψηλών ταχυτήτων και ιδίω στις σιδηροδρομικέ μεταφορές και έτσι πολλοί διαξιδιώτε προτιμούν ε, αυτές του ε, τους των ε, μεταφορών αντί για τα αεροπορικά ταξίδια, τρένα δηλαδή, αυτοκινητόδρομος, για τα ένα μεγάλη τα τρένα μεγάλης ταχύτητας. Είναι λοιπόν πιο πολύ οι, οι εταιρείε οι οποίες διαχειρίζονται τους σιδηροδρόμους και υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός για τις εταιρείε για να πάρουν τις άδειε ε, λειτουργίες και εκκριμένων γραμμών κλπ. Αυτά λοιπόν είναι καινούργιες εξελίξεις του τομέα. Και θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή τη νέα τάση, ας πούμε, και στο μέλλον και η τρίτη μου παρατήρηση, ερώτηση μάλλον, είναι αν η Κομισιόν είναι ευχαριστη... ικανοποιημένη με τις ε, εσωτερικές, ε, ε, με τα εσωτερικά ταξίδια, μέσα σε μια χώρα δηλαδή και όχι στο εξωτερικό. Εάν είναι ικανοποιημένη με Ε, τους ορισμούς που θα πρέπει να αποκλείουν αυτά τα, του είδους τα πακέτα ε, και αν πιστεύουν ότι ε, καλύπτεται αυτό το θέμα παρκώς των εσωτερικών μετακινήσεων. Εν συνεχεία τη δικαιοδοσία για τις ε, δια, υπερσυνοριακές μετακινήσεις και ταξίδια. Υπάρχουν αλλαγές στο νομικό κλίμα ειδικά αλλαγές που επήλθαν ε, με την οδηγία των δικαιωμάτων καταναλωτών. Εάν υπάρχουν ας πούμε νέες ε, διαδικασίες για αποζημιώσεις ε, σε περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων, διασυνοριακών ταξιδιών και επίση ευθύνε σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας ταξιδιωτικής εταιρείας που εδρεύει σε μια χώρα και των ταξιδιωτών που βρίσκονται στην άλλη χώρα. Ε, τα διασυνοριακά θέματα, χρεοκοπίες κλπ. Αυτά είχα να παρατηρήσω. Όχι ακόμα, άσε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και συγχαίρω και τον εισηγητή Είμαστε πολύ ευτυχείς που η ΙΜΚΟ αποφάσισε ένα σχετικά αυστηρό διάγραμμα. Αυτό δείχνει ότι προσδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα και πιστεύετε να ολοκληρωθεί το όλο θέμα και να έρθει στην Ολομέλεια στην, το Μάρτιο. Ε, θέλω να σας πω ότι όταν αναθεωρούμε τις προτάσεις ε, κάνουμε μία ευρεία ανασκόπηση και μελέτη του δικτύου προστασίας που υφίσταται σήμερα για τους ταξιδιώτες και τα δικαιώματά τους. Αν θυμόσετε το 1990 άρχισε η συζήτηση, δεν υπήρχε καθόλου στο παρελθόν. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν επιλογές σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο τμήμα εκείνο του ταξιδίου που, ε, που εμπλέκει τη μεταφορά, τη μεταφορά του ταξιδιώτη. Ε, αυτή, βασικά, αυτός βασικάς είναι ο στόχος μας και ε, ε, είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε περαιτέρω, διότι μπορούμε να φανταστούμε πολλές περιπτώσεις όπου είναι πολύ δύσκολο για έναν καταναλωτή να απευθυνθεί μόνο στον διοργανωτή ε, του ταξιδιού ή του πακέτου πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι δεν επιτρέπεται να λάβεις δύο αποζημιώσεις, διπλή αποζημίωση και από το ταξιδιωτικό μεταφορέα και από το ταξιδιωτικό γραφείο για την ίδια περίπτωση. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ένας ταξιδιώτης έχει αποζημιωθεί για μια καθυστέρηση, για μια ακύρωση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές ότι δεν πρέπει να καταβληθεί διπλή αποζημίωση σε αυτόν από δύο διαφορετικές πηγές. Πρέπει λοιπόν αυτό να είναι καθοριστικό. Το άλλο θέμα είναι να ευθυγραμμίσουμε τις δικές μας προτάσεις με την ε, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών όσον αφορά τον περιορισμό του αριθμού των διανυκτερεύσεων που πρέπει να καταβληθούν στον ταξιδιώτη από την αεροπορική εταιρεία σε περιπτώσεις ε, έκτακτης ανάγκης, ανατέρας βίας. Αριθμός των γενικτερεύσεων. Οι συνάδελφοι στην DG Move ε, συζητούν εις βάθος ε, αυτές τις νέες προσεγγίσεις και πρέπει να εξασφαλίσουμε συνέπεια, συνοχή στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Έχουμε επίσης διευκρινίσει και στην πρόταση και στην ανακοίνωση ότι η προσέγγιση μας βασίζεται όχι μόνο ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε όλα τα δικαιώματα στους ταξιδιώτες, αλλά και ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας. Ε, λόγω ενός συνδυασμού ε, των ταξιδιωτικών υπηρεσιών πρέπει να έχει και ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας. Τώρα σημείωσε την παρατήρηση που κάνετε για τις νέες εξελίξεις ε, τις, ε, στον ε, οδικό και σιδηροδρομικό τομέα μεταφορών. Θέλουμε οπωσδήποτε είναι διαλειτουργικό το, η νομοθετική αυτή πρόταση που εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές μεταφορών θα έχουμε την ευκαιρία στις συζητήσεις που θα κάνουμε να δούμε αν χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές σε συγκεκριμένες μορφές μεταφορών. Αλλά πιστεύουμε ότι, είπε όπως είπε και ο συνάδελφός μου, είχαμε μια πάρα πολύ μακρά διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους από όλους τους μεταφορικούς τομείς. Και δεν πιστεύω δεν μας ε, δεν μας είπαν ότι χρειάζεται να προσέξουμε ειδικά έναν τομέα περισσότερο από τους άλλους τομείς και έτσι τους αντιμετωπίζουμε διατομεακά. Ε, πρέπει επίσης να προσέξουμε ε, την αγορά αυτή οποία έχει ε, ιδιαιτερότητες ε, από πλευράς καταναλωτών. Υπάρχουν πολλές πτυχές που μπορούν να καλυφθούν από υπάρχουσα νομοθεσία, εφαρμοστέο δίκαιο, Ρώμη 1, συμβάσεις που ήδη υπάρχουν. Λάβαμε υπόψη και τη χάρτα για τα δικαιώματα του καταναλωτή Υπάρχουν τώρα καινούργιες απαιτήσει που υπάρχουν στην πρότασή μας βασίζονται λοιπόν σε αυτά τα νέα νομοθετικά μέσα, νέες νομοθετικές πράξεις για την προστασία των καταναλωτών και τέλος λάβαμε υπόψη και τα θέματα που άπτονται διασυνοριακών δραστηριοτήτων, όπως ας πούμε αν υπάρχει η χρεοκοπία μιας εταιρεία στο κράτος Α και τα σήματα στο κράτος Β κλπ πρέπει να βοηθήσουμε να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές ενέργειες και τη διασυνοριακή ε, αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έτσι Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε και δι με τη δική σας βοήθεια. Πρόεδρος, νομίζω ότι είναι ένας σαφής ε, στόχος αυτός και θα ακολουθήσουμε τη δική σας ηγεσία. Αναφέρθηκε και το χρονοδιάγραμμα και στις 4 ή 5 Νοεμβρίου έχουμε προγραμματίσει μια ακρόαση και πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα για να έχουμε ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας. Έτσι λοιπόν αυτό θα είναι μια πρόκληση για τον συγγετή και τους κοιόδες και θα συνεργαστούμε και με τη Μετροπή Μεταφορών. Θα διασφαλίσουμε λοιπόν ότι και τα δικά του συμφέροντα και απόψεις εκπροσωπούνται. Ανυπομονώ λοιπόν γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την Κομισιόν και όλη την ομάδα σας και ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε και να είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μέχρι του χρόνου το Μάρτιο. Λοιπόν, θα διακόψουμε για πολύ λίγο για να αλλάξει η ομάδα της Κομισιόν, γιατί έχουμε τώρα την ε, ομάδα από τη ΓΑΜΑ Είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό αυτό το απόγευμα για την Επιτροπή, γιατί συζητάμε δύο προτάσεις, όχι απλώς μία. Θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιους φίλους από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Connect, τον Ρομπέρτο Βιόλα και την ομάδα του και έχω τον προνόμιο να μου έχει ζητήσει η Επιτροπή να αναλάβω την ευθύνη για τρίτη φορά το πακέτο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας και που τα αφήνετε στα χέρια μου. Θα ήθελα να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ήμουν ε, ο εισηγητής για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες στο τελικό πακέτο. Το 2002 νομίζω συμφωνήθηκε ή τα Χριστούγεννα του 2001. Είχα χάσει ένα χρόνο, τέλο πάντων, έχει περάσει πολύ καιρό και επίσης ήμουν και εισηγητή αυτή τη επιτροπής για την μεταρρύθμιση αυτού του πακέτου που συμφωνήθηκε το 2009 και θα θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ ότι δεν καταρθώσαμε να συμφωνήσουμε στο τελικό πακέτο, ε, μάλλον καταρθώσαμε να συμφωνήσουμε στο τελικό πακέτο πριν από τις ευρωεκλογές στο Στρασβούργο και θα έλεγα ότι πάλι εδώ έχουμε μια νέα ενδιαφέρουσα πρόταση επιτάπητος και η κυρία Ρούλε και εγώ νομίζω έχουμε εργαστεί και στις δύο αυτές δεσμές μέτρων. Καλωσορίζω την κυρία Μπάστος ως νέο μέλος αυτής της ομάδας γιατί νομίζω ε, ε, ότι όσοι ήταν σκιώδεις στα προηγούμενα πακέτα θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Εσείς τώρα εδώ έρχεστε να συνεισφέρετε με νέες εμπειρίες και ιδέες. Αυτά για να πλαισίσω τη συζήτηση και να πω επίσης ότι έχουμε ήδη μία βασική συμφωνία με, με την Επιτροπή Βιομηχανίας ότι θα είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα τμήματα του πακέτου που αφορούν ε, τους χρήστες. Έτσι λοιπόν ε, θα δούμε και που θα επικεντρωθούμε σήμερα για τις τροπολογίες. Φυσικά οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες αν το επιθυμούν και για άλλα τμήματα του πακέτου, όμως εγώ θα έλεγα να επικεντρωθούμε το θέμα που αφορά τα δικαιώματα των χρηστών. Γιατί στο παρελθόν εγώ με την υποστήριξη της Επιτροπής ε, και διαπραγματεύτηκα με το Συμβούλιο είχα εισαγάγει κάποιες σημαντικές βελτιώσεις στα δικαιώματα των χρηστών και ξέρω ότι επεκτείνονται σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή τη νέα πρόταση και σημείωσα ότι έχουμε κάνει και πολύ καλή δουλειά για ε, τα ανώτατα όρια των ε, συμβολέων και ήταν ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόοδος που έγινε από αυτή την Επιτροπή. Όμως, τώρα ε, θα έχουμε διαθέσιμο και μία σύμβαση για 12 μηνών, δηλαδή θα περιοριστεί το χρονικό διάστημα, αλλά αυτή είναι μία λεπτομέρεια. Ξέρω ότι έχουμε αρκετή εμπειρία σε αυτό το τομέα και επίσης έχουμε και κάποια θέματα που αφορούν την περιαγωγή, το roaming. Και θα τα εξετάσουμε με την Επιτροπή Βιομηχανίας, γιατί πολλά από αυτά τα στοιχεία για την περαιτέρω μεταρρύθμιση του πακέτου περιεγωγής ε, δεν αφορούν ε, θέματα καταναλωτών, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα καταναλωτών και είναι πολύ σημαντικό να εισαχθούν κάποια μηνύματα προς τους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης για το κόστος της περιαγωγής και της περιαγωγής δεδομένων. Αυτά τα θέματα τα συζητούμε με την Επιτροπή Βιομηχανίας, έχουμε πολύ καλή σχέση με τους συναδέλφους από εκεί. Έτσι λοιπόν όλα αυτά για να κάνω μια εισαγωγή για το θέμα. Δεν ξέρω ποιος από την Κομισιόν ε, θα παρουσιάσει το θέμα αυτό, αλλά σίγουρα θα αναλύσουμε σήμερα το απόγευμα κάποια από τα στοιχεία που αφορούν ε, τους καταναλωτές προκειμένου να αποφασίσουν οι συνάδελφοι πώς θα προχωρήσουν με τις τροπολογίες, πώς θα κινηθούν σχετικά. Ρομπέρτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω και ο Άντων θα συνεχίσει με τη μελέτη αντικτύπων, συμφωνείτε. Η δική μου παρουσίαση είναι κατά κάποιο τρόπο μια εισαγωγή στο πακέτο. Επικεντρωνόμαστε στα στοιχεία που αφορούν τους καταναλωτές, αλλά αισθανθήκαμε ότι είναι χρήσιμο για την Επιτροπή να έχει μια ευρύτερη εισαγωγή για τη δέσμη μέτρων. Το πακέτο αποτελεί τμήμα της προσπάθειάς μας να επικεντρωθούμε στην ε, ε, αλλαγή, στην ε, μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια ψηφιακή οικονομία που έχει αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και αυτό αποτελεί τμήμα του ψηφιακού θεματολογίου. Δηλαδή αυτό το πακέτο δεν καλύπτει τα πάντα που αφορούν το ψηφιακό θεματολόγιο, αλλά έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα, με ένα τρόπο που να τα θέτει όλα μαζί και να αποτελεί το συγκολητικό στοιχείο, γιατί χωρίς ε, τη συνδεσιμότητα δεν έχουμε το υπολογιστικό νέφος, ούτε θα έχουμε πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών. Αυτό είναι το κύριο building block που χρειάζεται για μια συνδεδεμένη κοινωνία. Στις 10 Σεπτεμβρίου το Σώμα των Επιτρόπων υιοθέτησε ένα πακέτο που είναι το λεγόμενο Connected Continent, δηλαδή συνδεδεμένη ήπειρος και αποτελείται από τρία κυρία στοιχεία. Καταρχήν έχουμε μία ανακοίνωση που παρουσιάζει το όραμα της Κομισιόν για τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά στις τηλεπικοινωνίες. Και ο κανονισμός είναι πιθανότατα πιο σημαντικό βήμα για την πρόοδο, αλλά δεν είναι και το έσχατο. Η Κομισιόν έχει οθετήσει μία σύσταση για το κόστος και τιμή εισαγωγή διακρίσεων που σχετίζονται με το πρόσβαση στο βρυζανικό δίκτυο και πιθανότατα βλέπουμε την πρόσβαση της επόμενης ε, στα δίκτυα επόμενης γενιάς για να υπάρχει σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τις τιμές της πρόσβασης και εκεί επικεντρώνεται η σημερινή παρουσίαση και μια πρόταση κανονισμού που αφορά την ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών και φυσικά αυτό το πακέτο της συνδεδεμένης επίρου Connected Continent. Καταρχήν, γιατί κανονισμός. Αυτό είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να δούμε θέματα που σχετίζονται με τις καταναλωτές. Ο λόγος ε, για τον οποίο το νομοθέτημα του κανονισμού έχει επιλεχθεί είναι επειδή μιλάμε για την εσωτερική αγορά, δηλαδή μιλάμε για μέτρα εναρμόνισης και ως κάποιο βαθμό και σε ορισμένες περιπτώσεις μέγιστη εναρμόνιση. Επομένως, αναζητούμε παρόμοιες λύσεις παντού στην Ευρώπη και φυσικά ο κανονισμός είναι το κύριο νομοθέτημα που θα το πετύχει αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα που σχετίζεται με το χρόνο, με την ταχύτητα της εφαρμογής του όλου πακέτου. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε την οδηγία θα έπρεπε να έχουμε και ένα δεύτερο στάδιο της μεταφοράς της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και όλο αυτό θα καθυστερούσε την όλη διαδικασία της εφαρμογής. Η φιλοσοφία αυτού του πακέτου είναι ότι βασίζεται στο εφιστάμενο πακέτο και οικοδομεί πάνω σε αυτό και προσπαθεί να το συμπληρώσει και να το βελτιώσει εν ώψη μιας εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα. Το πακέτο αποτελείται βασικά από τρεις πυλώνες. Έχουμε ένα πρώτο πυλώνα που αφορά τον ενίο χώρο καταναλωτών, δηλαδή να πετύχουμε στο μέτρο του δυνατού τους ίδιους κανόνες, τις ε, ίδιες συνθήκες σύναψης συμβάσεων για τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη και φυσικά εδώ μιλάμε και για ε, συμβάσεις συνδεσιμότητας. Δεν μιλάμε για συμβάσεις που αναφέρονται στην αγορά υπηρεσιών και αγαθών στο διαδίκτυο. Στον πυλώνα αυτό έχουμε διατάξεις που αφορούν το ε, κλήσεις, δηλαδή τη διεθνή περιαγωγή και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο συσκευή του σε όλη την Ευρώπη και για τις διεθνείς κλήσεις. και στον πυλώνα των καταναλωτών για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουμε μία πρόταση για την ε, ουδετερότητα του δικτύου. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις εταιρείε, δηλαδή οι εταιρείε να μπορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη να προσφέρουν υπηρεσίες επικοινωνίας με τον πλούστερο δυνατό τρόπο. Και για μας ο πλούστερος δυνατός τρόπος είναι ότι πρέπει να κερδίσουν μια έγκριση, να λάβουν μια έγκριση και κατόπιν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άδεια αυτή που έχουν αποκτήσει ένα κράτο μέλο για να προσφέρουν υπηρεσίε σε όλα τα κράτη-μέλη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απλούστευση των προποθέσεων αδειοδότηση. Το τρίτο στοιχείο αφορά τι ουσιαστικέ ε, ε, συνεισφορές, τα input που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες για την προσφορά των υπηρεσιών. Έχουμε καταρχήν τα εικονικά προϊόντα, που είναι βασικά τα προϊόντα συνδεσιμότητας που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία για να οικοδομήσει μία προσφορά προς τους τελικούς καταναλωτές και οι συχνότητες, δηλαδή το φάσμα. Εδώ περιορίζουμε την προσοχή μας ε, ε, στο φάσμα, αλλά θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες όλους τους πολίτες ε, παντού στην Ευρώπη, όπου και αν βρίσκονται. Η ταχύτητα με την οποία οι υπηρεσίες ε, δεδομένων αυξάνονται στα κινητά είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει πάρα πολλές τέτοιες ε, προβολές και η επόμενη Κάθε φορά οι εξελίξεις ξεπερνούν την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν όλες οι συσκευέ μας σύντομα θα είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα τα αντικείμενα που θα είναι γύρω μας θα είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Επομένω, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επακές φάσμα για να καλύψουμε όλα όσα θα συμβούν σε μια συνδεδεμένη, υπερσυνδεδεμένη κοινωνία. Πολύ σύντομα θέλω να επικεντρωθώ στην πτυχή των καταναλωτών, γιατί καταρχήν είναι απαραίτητο να έχουμε ομοιομόρφους κανόνες ε, όταν ε, μιλάμε για την αγορά και τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Για, δύο, για ένα διτό λόγο. Καταρχήν, πρέπει να έχουμε το ίδιο επίπεδο προστασία σε όλη την Ευρώπη για να αποφύγουμε οι πελάτες σε ένα κράτος μέλος να είναι πιο προστατευμένοι από σε ένα άλλο. Γιατί αυτό δεν έχει νόημα σε μια νέα αγορά. Και όλος λόγος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε όταν ε, θέλουν να μπουν σε μια συγκεκριμένη αγορά να γνωρίζουν ε, ποια νομοθεσία πρέπει να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένη αγορά και αν αυτοί οι κανόνες την χάνει να είναι οι ίδιοι παντού τότε μπορούν ε, να κάνουν οικονομίες κλίμακας ε, και πεδίου ό,τι αφορά τις προσφορές. Πολλές φορές έχουμε εταιρείε ε, που μας λένε ότι για να αναπτύξουν και ιδιαίτερα εταιρείε που δραστηριοποιούνται σε πάνω μιας χώρας να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα για τους χρήστες ε, κοστίζει πάρα πολύ γιατί διαφέρουν οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Σήμερα έχουμε τεράστιες διαφορές παραδείγματος χάρη μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν ε, η προσφορά θα ήταν ίδια και θα επωφελούνταν και οι εταιρείε αλλά και οι καταναλωτές γιατί οι προσφορές θα είναι φτηνότερες. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που πιστεύουμε ότι είναι δικαίωμα του καταναλωτή είναι να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις ε, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας εντός της Ευρώπης σε μια λογική τιμή. Φυσικά η αγορά είναι αυτή που καθορίζει την τιμή, δεν γίνεται αυτό μέσω της νομοθεσίας, αλλά όταν ε, έχουμε ένα υπερβολικό κόστος που έρχεται από υπερβολικές τιμές περιεγωγές ή αδικαιολόγητες διαφορές στο κόστος των διεθνών κλήσεων, αυτό πρέπει να αρθεί, να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην εσωτερική αγορά. Ε, σήμερα, αν κάνουμε ένα τηλεφώνημα από τη Λισαβόνα στο Βίλνιους, παραδείγματος χάρη, αγορα σημερα αν κανουμε βιομηχανικά 3-4 λεπτά του ευρώ και υπάρχει και το κόστος έναρξης κλήσης και λήξης κλήσης που έχει μειωθεί σημαντικά, όμως παρόλα αυτά οι ταρίφες ε, που ισχύουν για το κοιμό μπορεί να είναι μέχρι και 1,5 ευρώ, όπως παίρνουμε το σχάρι πριν 20 χρόνια. σαν να μην ε, είχαμε όλη αυτή την απελευθέρωση και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Γι' αυτό βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά όποιοι και να είναι οι λόγοι, Νομίζω ότι είναι λογικό να αναμένουμε ότι στην εσωτερική αγορά αυτές οι διαφορέ μεταξύ του βιομηχανικού κόστους και της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτή θα πρέπει να συρρυκνωθούν σε κάποιο βαθμό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συμβάσεις, τα συμβολέα θα θέλαμε όλες οι προσυμβατικές πληροφορίες ε, που δίνονται στους καταναλωτές να είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θέλουμε εδώ μέγιστη εναρμόνιση των κανόνων. Αυτό για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και για να αποφύγουμε οι εθνικές αρχές να προβούν σε gold plating των ευρωπαϊκών κανόνων. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες για το τι προτείνουμε. Αλλά φυσικά αν υπάρξουν τέτοιες ερωτήσεις για αυτές ε, τις προ... για αυτά ε, τις προϋποθέσεις, για τους όρους που ισχύουν, πριν τη σύναψη του Συμβουλίου, ευχαρίστω να απαντήσω. Ένα άλλο θέμα που αφορά τους καταναλωτέ είναι το θέμα της διαφάνειας και των εργαλείων σύγκριση. Σήμερα Έχουμε αποδείξεις και θα τις παρουσιάσει ο συνάδελφος ότι δεν έχουμε εγκυμένη διαφάνεια στην Ευρώπη και οι ταχύτητες ε, που είναι αντικείμενο διαφήμισης δεν είναι αυτές που λαμβάνουν οι καταναλωτές, ούτε υπάρχει ενημέρωση για τις εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται ε, και σε πάρα πολλές δικαιοδοσίες δεν έχει δικαίωμα ο καταναλωτής να γνωρίζει. Εμείς πιστεύουμε βεβαίως στον ανταγωνισμό και στην ελεύθερη αγορά και ο καταναλωτής είναι το πρόσωπο κλειδί Δηλαδή αυτός θα πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις αλλά θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι ελεύθερος να αποφασίσει για το καλύτερο. Τώρα, ουδετερότητα του δικτύου, σημαντικό στοιχείο της πρότασης αυτής. Είναι η πρώτη φορά που στο ευρωπαϊκό κεκτημένο υπάρχει μία πρόταση να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό. Και αν ε, θεωρήσουμε ότι η ιστορική μας αγορά έχει ένα εκατομμύριο πολίτες, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη προσπάθεια στον κόσμο για να νομοθετήσουμε στην ουδετερότητα του δικτύου. Να σας υπενθυμίσω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν πραγματική νομοθεσία γιατί η FCC απεφάνθη για την ε, ουδετερότητα του δικτύου και τελικά ποτέ δεν κατέληξε όλο αυτό σε νομοθεσία. Έτσι λοιπόν, η Κομισιόν θεωρεί ότι καθώς έχει το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, σκέφτηκε ότι ο πιο δημοκρατικός τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου είναι να έχουμε νομοθεσία. Φυσικά όχι να παρεμποδίσουμε τις εξελίξεις, αλλά να έχουμε ένα ελάχιστο σύνολο αρχών. Και προσπαθήσαμε την οδό των συστάσεων, αλλά κατόπιν οι νομικοί εμπειρογνωμές μας είπαν ότι αν δώσουμε εξουσίες στις NRAs για να ε, μπλοκάρουν παραδείγματο χάρη κάποια τμήματα, δεν θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο για ε, να γίνει χωρίς νομοθεσία. Έτσι λοιπόν η νομοθεσία αφορά τις ελάχιστες εγγύησεις που θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε πελάτη και αυτό αποτελεί ότι έχουμε ανοιχτό ίντερνετ και αυτό υπερισχύει, δεν υπάρχει μπλοκάρισμα των σελίδων και θα πρέπει διαχείριση της κυκλοφορίας να γίνεται χωρίς εισαγωγή διακρίσεων. Αυτή είναι και οι κυρίες αρχές, την πρότασή μας για την ιδιαιτερότητα του δικτύου και επιτρέπουμε κάποια καινοτομία σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες, γιατί επιτρέπουμε να προσφέρονται και ειδικέ υπηρεσίες υπό τον έλεγχο των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιαγωγή, αφού έχουν περάσει κάποιοι μήνες από την ε, έγκριση του Roaming 3 θα αναρωτηθείτε γιατί επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε τώρα από μια σκοπιά εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι ένας λόγος. Ο λόγος είναι ότι στο πακέτο αυτό, ας το αποκαλέσουμε roaming, η περιεγωγή 4, είναι ένα εθελοντικό καθεστώς. Δεν αλλάζει δηλαδή το roaming 3, αλλά προσφέρει μια δυνατότητα, μια επιλογή στις εταιρείες να πούν το εξή. Αν ε, θα θέλετε να σκεφτείτε να προσφέρετε στις υπηρεσίες σας αυτή την επιλογή μέσω συμμαχιών ή συμφωνιών ή μέσω ενός εναλλακτικού παρόχου, τότε μπορεί να απαλλαχθείτε από κάποιες από τις υποχρεώσεις στο roaming 3. Και γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό ταιριάζει με την εσωτερική αγορά, επειδή τελικά συμπεριλαμβάνει εδώ και καλύπτει τι εταιρείε που θέλουν να έχουν ευρωπαϊκή δραστηριότητα και επίσης αλλάζει και κάπως το παράδειγμα στην περιαγωγή. Γιατί η τελική περιαγωγή μπορεί να γίνει αν οι εταιρείε μπορούν να εσωτερικεύσουν το κόστος. Γιατί αν κάνεις περιαγωγή εκτός ε, του εσωτερικού σου δικτύου ή των ε, συμμάχων σου, τότε πάντοτε θα είναι εξωτερικό το κόστος. Ποτέ λοιπόν δεν μπορεί να είναι μηδενικό το κόστος, γιατί ουσιαστικά βγαίνει εκτός του δικτύου. Αν αντίθετα είναι εντός του δικτύου ο πελάτης, και εδώ μιλάμε για ένα ευρύτερο δίκτυο που περιλαμβάνει και τις συμμαχίες, τότε μπορεί να εσωτερικευτεί το κόστος και πιστεύουμε ότι μπορεί να αντισταθμιστεί περισσότερο ή 100%. Έτσι λοιπόν εισαγάγοντας σταδιακά αυτή τη δυνατότητα με την εσωτερικοποίηση του κόστος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε κανένα δύο χρόνια μπορούμε να εξελίψουμε την περιαγωγή. Και από όταν θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό ο κανονισμό προτείνουμε να μην υπάρχει χρέωση για την εισερχόμενη κλίση που σήμερα πραγματικά σε μεγάλο βαθμό δεν δικαιολογείται γιατί έχουμε τον τερματισμό ε, της κλίσης που ήταν ως πριν και έχει τώρα καταληφθεί. Τώρα, θα σταματήσω εδώ, επειδή βλέπω και να περνάει η ώρα. Έχουμε τώρα και άλλα σημεία που αφορούν την ενιαία έγκριση, το φάσμα που είναι λιγότερο σχετικά και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ναι, νομίζω ότι αναφέρατε τα βασικά στοιχεία που θα εξετάσουμε και ξέρουμε τώρα ποιε ερωτήσει πρέπει να θέσουμε σήμερα το απόγευμα. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας μιλήσω για τη διαφάνεια που έχει να κάνει με τους στόχους της πρότασης αυτής. Να, θέλω να βρω τη σωστή διαφάνεια, συγγνώμη δύο λόγια για αυτή τη διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων. Είναι σημαντική αυτή η αξία. Ένα από τα σημεία εκκίνησης για την αξιολόγησή μας ήταν η αίσθηση του επίγοντος που είχαμε. Πρέπει ο τομέας να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο ύψος των προκλήσεων, των ετοιμάτων που, ε, που ε, διατυπώνει η ευρύτερη κοινωνία αλλά και η οικονομία αν θέλετε. Και γι' αυτό δεν κάναμε συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση, αλλά ε, είχαμε πολύ ευρείες επαφές με πολλούς και διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα κράτη-μέλη. Έγινε μια πολύ εκτεταμένη δουλειά από τον Πάρικ συμπεριλαμβανομένου και του θέματος του ανοιχτού ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένου των θεμάτων για τη διαφάνεια. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και εύγλωτα σε σχέση και με το IRSPG Είχαμε πολλές συναντήσεις με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο σε μια δημόσια συνεδρίαση τον Ιούνιο, εκτός από πέρα, εκτός από τις, και πέρα από τις δικές μας δραστηριότητες, όπου πάντοτε βεβαίως μελετούμε, συλλέγουμε στοιχεία, αξιολογούμε και το καθεξής. Είναι ένα μέτρο λοιπόν εσωτερικής αγοράς και δεν θα πρέπει να σας εκπλήξει αυτό το γεγονός. Ο κατακαιρματισμός της αγοράς είναι ο κοινός τόπος που έρχεται στο προσκήνιο ξανά και ξανά ε, για θέματα φάσματος, για θέματα πρόσβασης σε δίκτυα. Και κάτι που είναι πιο σημαντικό εδώ, για θέματα προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή, ο κατακαιρματισμός είναι το βασικό χαρακτηριστικό τεράστιος και ευρύς κατακαιρματισμός στις κανονιστικές προσεγγίσεις, στις νομοθετικές προσεγγίσεις σε κάθε χώρα, ακόμα και έχοντας τη βάση των ελάχιστων προτύπων ή προδιαγραφών ε, των υφιστάμενων οδηγιών. Παρόλα τα αυτό ο κατακαιρματισμός παραμένει και αυτός ο κατακαιρματισμός είναι που έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις ε, για όλους τους εμπλεκόμενους και για τους καταναλωτές βέβαια πολύ μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές στις διάφορες αγορές τις ευρωπαϊκές και αυτό δεν εξηγείται από αντικειμενικές διαφορές στο κόστος εργασίας ή ε, σημαντικές διαφορές στη διαθεσιμότητα φάσματος για σύρματες υπηρεσίες. Το σημαντικό να πω ότι είναι το εξής. Η ανάλυση δείχνει ότι είναι τεράστιες οι αποκλήσεις στις τιμές. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η αύξηση της πρόσβασης θα οδηγήσει σε σύγκληση, ότι οι τιμές των φτηνών χωρών θα ανέβουν και οι, τιμές των, ε, οι ακριβές τιμές των χωρών των άλλων θα πέσουν. Θα, υπάρξουν, ε, θα υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση ως προς τις βέλτιστες πρακτικές των ανταγωνισμών. Εκεί όπου οι επενδύσεις είναι υψηλότερες, τα καλύτερα δίκτυα οδηγούν σε περισσότερη αποτελεσματικότητα, μείωση του κόστους και μετακύληση των πλεονεκτημάτων αυτών ε, στον τελικό χρήστη. Τρόπους λοιπόν να αντισταθμιστεί η, η απόκληση των τιμών είναι το γεγονός ότι ε, είναι διαφορετικές οι επιδόσεις στον κλάδο. Προσπαθεί η κάθε εταιρεία να, να προστατεύσει τη δική της θέση στην τοπική ή εθνική αγορά και δεν έχει το δυναμισμό να είναι πιο εξωστρεφής και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αυξανόμενης ζήτησης. διότι μια πιο ευρεία οικονομία εξαρτάται από μεγαλύτερη ε, διασύνδεση. Αυτό είναι σαφές. Βεβαίως εξετάσαμε την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της, ανατολικο... της αναλογικότητας και η παρέμβασή μας είναι η ελάχιστη δυνατή για να μειώσουμε στο ελάχιστο την παρέμβασή μας ε, πάνω σε θέματα για τα οποία δικαιολογείται εθνική αυτονομία ή περιφερειακή αυτονομία. Για παράδειγμα, δεν ασχολούμαστε καθόλου με τα αντισταθμιστικά μέτρα τα αντισταθμιστικά ωφέλη για τη χρήση του φάσματος. Δεν προτείνουμε μια νέα ρυθμιστική αρχή, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι ε, σοφρόνος πράττοντες έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές θα εντοπίσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό και τα, ο τρόπος να αντισταθμιστούν αυτά και η Κομισιόν θα βρει τρόπους να προωθήσει τη σύγκληση. Τώρα, ως προς την αξιολόγηση αντικτύπου, ε, πώς δομείται. Έχουμε τέσσερα σετ στόχων που ανταποκρίνονται σε τέσσερις ευρύς τομείς δράσης. Παροχή υπηρεσιών όσο ήταν τον πιο ενιαία, καθεστώς αδειοδότησης, μεγαλύτερη συνέπεια στο φάσμα, στην ε, ευρωπαϊκή χονδρική στα σταθερά δίκτυα και τη συνεισφορά της, στην προστασία του τελικού χρήστη. Και έχουμε και την προστασία των καταναλωτών ε, όταν ε, βρίσκονται σε διεθνή περιαγωγή. Επομένως, προσπαθώντας να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, πάλι εξετάσαμε ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές μας διαβάθμιση, σταδιακή προσέγγιση και διάνυση όλων αυτών των διαφορετικών δρόμων εν ώψη των διαφορετικών κανονισμών και βάση των διαφορετικών κανονισμών και οδηγιών, πρώτον. Δεύτερη επιλογή, ενιαίο νομοθετικό μέτρο, όχι πλήρη αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, συνδυασμός εστιασμένων παρεμβάσεων. Τρίτη επιλογή, να ακολουθήσουμε τη δεύτερη επιλογή και εκεί να προσθέσουμε περισσότερη κεντρική διαχείριση. Ε, περισσότερη ευρωπαϊκή κανονιστική εξουσία σε κεντρικό επίπεδο. Βεβαίως όλα αυτά είναι και θέματα εσωτερικών συζητήσεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, ως προς το ωφέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε ποιο αποτέλεσμα θα είχε η σύγκληση στις ευρωπαϊκές αγορές προς τις βέλτιστες ευρωπαϊκές αγορές και μιλώ κυρίως για τις τιμές. Και βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικά ωφέλη της άξης των δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Βεβαίως υπάρχουν και λιγότερο μετρήσιμα ωφέλη για τον ίδιο το κλάδο. Και περιλαμβάνεται και ο δημόσιος τομέας εκεί που θα ωφεληθεί από μια πιο υγιή αγορά με μεγαλύτερη και περισσότερη διασύνδεση. Συμπεριλαμβάνονται και οι τελικοί χρήστε. Δεν θα έχουμε μόνο την επίσημη βεβαίως προστασία κατοχήριωση των δικαιωμάτων τους ε, βάσει του κανονισμού, αλλά θα ωφεληθούν από, τον ε, από τη μεγαλύτερη ε, και πιο δυναμική ανταγωνιστικότητα. Το θέμα του κόστους τώρα. Εδώ εξετάσαμε τα χειρότερα δυνατά σενάρια και μάλιστα ευελεχώς για να έχουμε πλήρη συνέστηση αυτών που προτείνουμε. Είναι συγκεκριμένες διατάξεις που έχουν επίπτωση στα εισοδήματα, στα έσοδα των παρόχων Ωστόσο, για διάφορους λόγους πράγματι πιστεύουμε ότι το χειρότερο δυνατό σενάριο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, είτε διότι θα αυξηθεί η ζήτηση, θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, είτε γιατί είναι απαξιωμένα αυτά τα ε, επιχειρησιακά μοντέλα και αυτό είναι ευρέως αποδεκτό, άρα το μόνο που θα κάνουμε είναι να επιταχύνουμε ε, τις προαναγγελθήσεις εξελίξεις, είτε γιατί δεν θα πάμε προς, την, προς τον κανονισμό σκληρών, αν θέλετε, άκαμπτων τιμών, αλλά θα πάμε προς το να ενθαρρύνουμε πιο βιώσιμες πρακτικές. Σε, αυτό το, σε αυτή τη γραφική παράσταση βλέπετε την αξιολόγηση του συνολικού αντικτύπου και εξάγουμε κατά συνέπεια το εξής συμπέρασμα ότι η επιλογή υπαριθμών 2 είναι προτιμητέα, είναι προτιμότερη. Χωρίς να σας διαβάσω όλο αυτό το κείμενο της διαφάνειας, γιατί είναι πολύ πυκνό, το θέμα είναι ποιο πεδίο εφαρμογής θα έχει αυτή η δράση και σε ποιο βάθος χρόνου. Εάν εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια κανονιστική ε, πρόταση, τότε θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, γιατί μιλούμε για κανονισμό που θα αμέσως θα αρχίσει να ισχύει και να, να εφαρμόζεται. Πρέπει να επιτύχουμε τον στόχο της εναρμόνισης όλων αυτών που προτείνονται στον τελικό χρήστη. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε γρήγορη δράση και γρήγορη αντίδραση από τους λήπτες, από αυτούς που θα μπουν σε αυτό το καθεστώς και έχουμε ένα επαρκές πεδίο εφαρμογής ε, μέσα στο οποίο πράγματι θα επιληθούν τα πιο επίγοντα προβλήματα τα οποία ε, χρήζουν λύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος, καλώς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Well, I think it be useful. Ξέρω ότι είχατε πολλές συζητήσεις στην Επιτροπή Βιομηχανίας και δεν θέλω να τις επαναλάβω, να σχολιάσω τις συζητήσεις σας και τη φύση της ε, μελέτης ε, αντικτύπου. Όλα αυτά πολύ χρήσιμα, αλλά εμείς θέλουμε να προσέξουμε βασικά τις, ε, την πτυχή των καταναλωτών. Κυρία Μπάστος, έχετε τίποτα εσείς να προσθέσετε. Σας πειράζει αν εγώ ρωτήσω θέσω ορισμένε ερωτήσεις πρώτα ή θέλετε να προηγηθείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, αυτής της ε, σημαντικής έκθεσης. Πιθανότατα η δική μου παρέμβαση θα είναι κάπως κατά αυτού του ρεύματο ενθουσιασμού που είναι εμφανής ε, εδώ από την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά αυτή ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μια μελέτη η οποία αιτιολογεί την υιοθέτηση νομοθεσία. Είναι σπάνιε οι φορέ που κάτι τέτοιο συμβαίνει σε αυτό το κοινοβούλιο, να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιοι είναι οι λόγοι που ουσιαστικά βρίσκονται στην πηγή της απόφασης για νομοθέτηση. Εγώ ελπίζω ότι αυτή η οδός που ξεκινά σήμερα να μας οδηγήσει σε μια ισορροπημένη κατάσταση ε, και να καταπολεμήσουμε το γεγονός ότι νομοθετούμε άσχημα και υπερβολικά. Τώρα εδώ θέλουμε να ξέρουμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε παρκώς σχετικά με την ευκαιρία αυτής της νομοθεσίας ακόμη και υπό την οπτική της προστασίας ε, του καταναλωτή. Εγώ έχω κάποιες συμφιβολίες γιατί υπάρχουν πολιτικές, νομικές και οικονομικές επιπτώσεις στο θέμα αυτό. Από πολιτική σκοπιά φαίνεται πως η πρόταση αυτή παρόλο που είναι αξιέπαινη η προσπάθεια αυτά έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Βρισκόμαστε στο τέλος θητείας μας και σε προεκλογικό πλαίσιο και πολλές ε, φορές αυτό δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε λογικά και ισορροπημένα και επίση αυτό το χρονοδιάγραμμα μας θέτει ένα χρονοδιάγραμμα ασύμβατο με τη συζήτηση αυτή. Αυτό το θέμα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πρέπει να το λάβουμε υπόψη και επίση, η ουδετερότητα του δικτύου πέρα από ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τα μάλα και επειδή μας απασχολεί τα μάλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με πολύ μεγάλη ευαισθησία γιατί μιλάμε για θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία της έκφρασης, της παροχής υπηρεσιών, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και φυσικά θίγονται δικαιώματα που θεωρούμε ότι είναι πιο καθολικά και δεν θα έπρεπε εδώ να υπάρχουν δημαγωγικές και λαϊκιστικές προσεγγίσεις. Δεν ήταν ξεκάθαρο για μένα κατόπιν ε, της ανάγνωσης αλλά και των συνεισφορών που ξέρουμε, ποια είναι η καλύτερη χρονική στιγμή για την υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας από νομική σκοπιά. Αυτή η πρόταση κανονισμού σχεδόν ε, αναθεωρεί όλη την ισχύουσα νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ορισμένα από τα θέματα αυτά ε, τέθηκαν σε ισχύ μόλις πριν λίγους μήνες. Ούτε καν τα κράτη-μέλη είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν την ε, νομοθεσία αυτή στο εσωτερικό τους δίκαιο. Επίσης κάτι που δεν, ε, που δεν είναι σαφές είναι για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάλεξε έναν νέο κανονισμό για να θεωρήσει διάφορες ισχύουσες οδικίες για τόσο διαφοροποιημένα ζητήματα όπως είναι η καθολική υπηρεσία, το roaming, δεύτερο το, το δικτύου κτλ. Και τώρα εγώ ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ βέβαια το Γενικό Διευθυντή και όλη την ομάδα. Τους ευχαριστώ για την παρουσίασή τους, αλλά θέλω να ρωτήσω μήπως θα ήταν καλύτερο να γίνει μια αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ακόμη και αν ε, είναι σε πρώιμο στάδιο, γιατί είναι σε ισχύ πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αντί να τίθενται κάποια τόσο ελκυστικά θέματα στο πακέτο από οικονομική σκοπιά. Εδώ μιλάμε ότι το κύριο ενδιαφέρον μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Αυτό μας απασχολεί σε αυτή την Επιτροπή. Σήμερα ισχύει ένα μια πολύπλοκη ε, τάξη που προσφέρει ασφάλεια δικαίου σε όλους ε, τους ε, πρωταγωνιστές και μιλώ και για τις εταιρείες και τις πιο μικρές τις ε, μεγαλύτερες αλλά και σε εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ και στους καταναλωτές. Και αυτή η ασφάλεια δικαίου είναι πολύ σημαντική για να έχουμε ένα θετικό επενδυτικό κλίμα, ανταγωνιστική αγορά και να γίνονται επενδύσεις στις υποδομές των τηλεπικοινωνιών. Όλα αυτά πάντοτε ωφελούν τα πολλά εκατομμύρια καταναλωτών που έχουμε στην Ευρώπη. Όμως σε μια συγκυρία κρίσης και δεν έχουμε βγει ακόμη από αυτή, ακόμη και αν ε, είμαστε αισιόδοξοι, η Κομισιόν αποφάσισε να αλλάξει εις βάθος τους ισχύοντες κανόνες σε ένα τομέα, σε ένα κλάδο που συνέχιζε να μεγενθύνεται. Και για να αναφερθώ συγκεκριμένα στο παράδειγμα της περιαγωγής που προκαλεί τι μεγαλύτερε εντυπωσει και μας αφορά περισσότερο σε αυτή την Κομισιόν. Η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία ευθύθηκε πριν ένα χρόνο, το 2012 και τότε ήδη είχε παρουσιαστεί ω μια νομοθεσία που προλάμβανε τις μελλοντικέ εξελίξεις στην αγορά και στην τεχνολογία. Τελικά αυτή η νομοθεσία δεν διήρκεσε ούτε κανένα μισή χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ πρόσφατες επενδύσεις τελικά διακυβεύονται από τη νέα πρόταση, η οποία τελικά είναι κατά οποιασδήποτε ιδέας προόβλεψης για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα μεταξύ όλων των παρόχων και των καταναλωτών. Και επίσης για αυτή την οικονομική προοπτική δεν ε, κατανοούμε ποιοι είναι οι λόγοι που παρουσιάζεται τώρα αυτή η πρόταση. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους που ανέφερα υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή του λόγου. Αναφερθήκατε ε, στο να δοθούν κίνητρα στην αγορά, να δοθεί όθηση στην αγορά και εμείς ε, σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές ε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όσο μεγαλύτερη δυνατότητα και ελευθερία επιλογής έχουν τόσο περισσότερο κερδίζει ο καταναλωτής. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προωθεί ευρωπαϊκούς γίγοντες για να ανταγωνιστούν στην παγκοσμία αγορά. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ο λόγος και Αυτά, το παράδειγμα που μας παρουσιάστηκαν δύο φορές ε, απερίφθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν υπήρχε επαρκής διδιολόγηση. Επίσης, η αξιολόγηση της μελέτης αντικτύπου δεν ήταν ε, πληρής, δηλαδή δεν ήταν το θετική το αρνητική. Και αυτό δημιουργεί νόμιμες εμφιβολίες για την αξιολόγηση που οδήγησε στην εκπόνηση αυτής της πρότασης. Όμως θέλω να κλείσω με κάτι θετικό παρά τις αμφιβολίες που επεσήμανα, είναι πολύ σαφές για τη δική μου ομάδα, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι αυτή είναι μία πρόταση η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά από εμά και εις βάθος. Και είμαι σίγουρη ότι σε συνεργασία με τον πρόεδρο Χάρμπουρ και εισηγητή της ΣΥΜΚΟ για αυτή τη σημαντική πρόταση θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που να είναι συνεκτικό και να προστατεύει τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much. Ευχαριστώ και εγώ. Λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω ότι αυτά τα επιχειρήματα ε, ακούστηκαν και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και μάλιστα έντονα. Το θέμα είναι ότι η πρόταση δεν θα μπορέσει να περάσει από το κανονιστικό σύστημα ως έχει σήμερα. Από πλευράς καταναλωτών θα ήθελα να ξέρω πρώτον και παρόλο που γνωρίζω το κεφάλαιο αυτό γιατί το έχω διαβάσει εις βάθος μου φαίνεται περίεργο να αντιγράφουμε ορισμένα σημεία της υπάρχουσας οδηγίας με ορισμένες επιπλέον διατάξεις. Και να το παρουσιάζουμε τώρα ως κανονισμό όταν ήδη έχουμε ένα κανονιστικό μηχανισμό όπου όλοι οι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν έχω δει λοιπόν μία αντίστοιχη μελέτη αντικτύπου και κάθε ανάλυση θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα τα, τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν ακόμα στα κράτη-μέλη και γιατί αυτές οι αδυναμίες, αυτές οι ελλείψεις θεωρούνται τόσο σοβαρές ώστε να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ευρωστία του τομέα. Δεν έχω διαπιστώσει κανέναν συσχετισμό, μεταξύ αυτού και της ανάπτυξης του τομέα ούτε έχω δει καμία αναφορά μεταξύ αυτής της ε, κατάστασης και της ε, όθησης νέων επενδύσεων από πλευράς της Επιτροπής μας θα ε, θεωρούσαμε πραγματικά ε, θα κάναμε μια ενημέρωση, μια επικαιροποίηση των κανονισμών ευχαρίστως εάν βοηθήσει την ε, υπάρχουσα οδηγία και την εφαρμογή της. Μερικές ένας εξυγχρονισμός θα μπορούσε να γίνει με κατευθυντήριες γραμμές και αυτό θα επιτάχυνε τη διαδικασία. Είμαι ευχαριστημένος που έχετε ενσωματώσει ορισμένε από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου μετά από την αρχική σας πρόταση αλλά το ότι αυτή τη στιγμή εδώ παρουσιάζεται κάτι το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τα ωφέλη προς τους ε, καταναλωτές, θα τα διευρύνει, θα τα ενδυναμώσει, δεν με πείθει. Ε, μου φαίνεται ότι η μεγάλη αδυναμία αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν είχαμε καμία ε, πρώτερη διαβούλευση ε, για το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είχαμε μία προηγούμενη ε, διαβούλευση πριν καταγράψουμε αυτές τις σημαντικές ελλείψεις για τις οποίες χρειάζεται όλη αυτή η αναθεώρηση. Καταρχάς μας ενδιαφέρει και ρωτώ τον Ρομπέρτο ειδικά και τον Άντωνη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τίτλος, οι επικεφαλίδες. Ότι πρέπει να επέλθει μία δικτυακή ουδατερότητα. Σε αυτή την οδηγία το θέμα της ε, δικτυακής ε, ουδετερότητος δεν αναφέρεται πουθενά. Ούτε καν υπάρχει στους ορισμούς αυτή η διαδικτυακή ουδετερότητα. Ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν αυτού, αυτής της πτυχής, γιατί αναφέρεται εδώ ποιος είναι ο λόγος. Εμείς εργαστήκαμε πολύ σκληρά στην αρχική οδηγία για την δρέωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Κατά πόσο λοιπόν πιστεύετε ότι υπάρχει ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα με το αντιανταγωνιστικό blocking για, που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Η έκθεση Μπέρεκ που είδα εγώ, που μελέτησα εγώ, αντιμετωπίζει ήδη αυτό το θέμα τα κατά του ανταγωνισμού. Μου φαίνεται ότι εσείς εισάγετε ορισμένα νέα στοιχεία στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών και μάλιστα νέους ορισμούς που δεν έχουν ανακύψει ποτέ στο παρελθόν. Ποιες είναι αυτές οι specialized services, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και ε, ε, τι σώοι προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα κενοφανή στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να καλύψει η υπάρχουσα οδηγία. Εφόσον λοιπόν μας ζητάτε να μελετήσουμε θέματα και ζητήματα τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσιών για τον τελικό χρήστη, πρέπει να καταλάβουμε ε, και γιατί ακριβώς πιστεύετε ότι προέκυψαν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας ε, μέχρι ως εδώ. Και ποια είναι αυτά τα νέα συνταρακτικά στοιχεία που έχουν προκύψει που μας αναγκάζουν να αναμορφώσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η πρώτη μας αντίδραση μαζί με τον Άντωνη ε, βεβαίως θα μπορέσουμε να εργαστούμε μαζί για να σας δώσουμε τα στοιχεία που χρειάζεστε και για τη δική σας εργασία. Αλλά εδώ είναι μια πρώτη αντίδραση. Δύο ζητήματα από υψηλά ιστάμενους πιστεύω ότι δεν παρουσιάστηκαν αρκετά ευκρινώς. Θέλουμε αυτός ο κανονισμός να ακολουθήσει μια εντελώς καινούργια οδό από ό,τι στο παρελθόν. Εμείς ε, θέλουμε να επιτύχουμε μια μέγιστη εναρμόνιση που είναι ε, μια εντελώς νέα κατεύθυνση από το παρελθόν. Λέμε λοιπόν ότι οι καταναλωτές, στα κράτη-μέλη α, β, γ δεν θα πρέπει να ωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο από καταναλωτές στα άλλα κράτη-μέλη. Διότι δεν βλέπουμε κανένα λόγο γιατί οι διαδικτυακές υπηρεσίες ε, και δι της προστασίας των καταναλωτών ε, πρέπει να είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και δεύτερον εταιρείε που επενδύουν από, μια, από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο πρέπει να αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Μιλάμε εδώ για προτυποποίηση. Προτυποποίηση λοιπόν και εναρμόνιση. Γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνουμε ορισμένα από τα στοιχεία που υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή παίρνουμε τα θετικά, τα καλά στοιχεία από το παρελθόν και ξέρουμε πόσο σημαντική ήταν η εργασία αυτή τη επιτροπή για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Παίρνουμε λοιπόν αυτά τα καλά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουμε στα, στις πρότυπες συμβάσεις. Στη μελέτη αντικτύπου υπάρχουν πάρα πολλά ε, πάρα πολλές ενδείξεις, στοιχεία που δείχνουν τις διαφορές στην Ευρώπη. Δημοσιεύσαμε μία μελέτη για τη διαφάνεια που ανατέθηκε στην εταιρεία Samnows και η ταχύτητα με την οποία διαφημίστηκε, η, η ταχύτητα η που διαφημίστηκε για τους καταναλωτές δεν είναι η ταχύτητα την οποία τελικά λαμβάνουν Επίσης, 300 εκατομμύρια πολίτες αυτή τη στιγμή μπλοκάρονται όταν ε, χρησιμοποιούν το Voice over IP. Τρία χρόνια συζητούμε λοιπόν ε, το θέμα της παροχής αυτών των υπηρεσιών και διαπιστώνουμε μία συλλογική ε, δεν υπάρχει μια συλλογική αποτυχία, αλλά ε, εν μέρη ορισμένα πράγματα έχουν αποτύχει και δεν υπάρχει και μια σταθερή βάση στην οποία μπορούμε να λειτουργήσουμε για να εφαρμόσουμε τα μέτρα κατά του μπλοκαρίσματος. Δεν υπάρχει δηλαδή επαρκής νομική βάση για να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε μία πρακτική η οποία είναι κατά του ανταγωνισμού, η οποία υπονομεύει τον ανταγωνισμό. έχετε δίκιο ότι σε ορισμένα μέρη επαναλαμβάνουμε τα, τα παρελθόντα σε αυτόν τον κανονισμό, αλλά και εμείς πρέπει να βασιστούμε στα χρόνια της εμπειρίας που έχουμε συλλέξει. Είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα όλος ο τομέας και τον ε, παρακολουθούμε πολύ αυστηρά την όλη σύνταξη της έκθεσης αντικτύπου. Ε, δεν βλέπω λοιπόν ε, ειλικρινά γιατί δεν είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους ζητούμε δράση. Βεβαίως, χρειάζεται περαιτέρω διαβούλευση με την Επιτροπή σας, εάν νομίζετε ότι λείπουν στοιχεία και αν μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερη στοιχεία και να σας καλύτερα, παρακαλώ πέστε μου το. Ε, ε, ε, εάν το επιτρέπει ο χρόνος, θα προσπαθήσω να σχολιάσω κάποια από τα βασικά σημεία για το ανοιχτό διαδικτύο, για την περιαγωγή και για το γενικότερο ε, τελικό χρήση και το μπλοκ των διατάξεων. Παίρνω το νήμα της συζήτησης από εκεί που το άφησε ο Ρομπέρτο για τις διατάξεις για το ανοιχτό διαδίκτυο. Είναι ένας τομέας όπου Είχαμε το όφελος της κλασικής τρίμηνης διαβούλευσης, λάβαμε εκατοντάδες απαντήσεις. Επομένως, τα στοιχεία που συλλέξαμε μετά από αυτή τη διαδικασία είναι αρκετά στέρεα. Πράγματι, δεν χρησιμοποιείται ο όρος ουδετερότητα στο νομικό κείμενο, ακριβώς διότι ο όρος αυτός, η έκφραση αυτή, έχει ε, φέρνει συνειρμούς στο πολιτικό επίπεδο που μας δυσκολεύουν κάπως. Θέλουμε να διατυπώνουμε νομοθετικές διατάξεις με βάση την προσέγγιση ε, επί των αρχών και θέλουμε να καλύψουμε νομικά κενά ε, βάσει της συμβουλής των δικών μας νομικών υπηρεσιών μετά από το άρθρο 3,1 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και το άρθρο 23, δηλαδή συνδυαστικά αυτά τα δύο. Μιλήσατε για την έννοια των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, είναι σημαντικό για να πετύχουμε δύο πράγματα που και αυτά έχουμε, έχουν σημασία. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο που θα ορίσουμε ε, θα είναι μια πρόσβαση που θα περιλαμβάνει τη μη διάκριση και το μη μπλοκάρισμα αν θέλετε, το, τη μη φραγή. Ε, και θα πρέπει αυτά τα δύο τελευταία να λέγονται κατάφορα και να είναι πολύ καλά προστατευμένα. Και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των παρόχων εφαρμογών θα πρέπει να υπάρχει ε, συμφωνία και ξεκαθάρισμα χωρίς να επιμολύνουν οι μεν τους δε και αντιστρόφως. Και όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν για να θεσπιστεί αυτή η νέα, να ενσωματωθεί αυτή η νέα νομική έννοια. Τώρα, ως προς το, την περιαγωγή, τον κανονισμό για την περιαγωγή που πρόσφατα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Μπάστος, έχουμε διάφορες διατάξεις. Ε, έχουμε πάρει τις διατάξεις αυτού του κανονισμού και τους έχουμε, τις έχουμε περιλάβει, άθικτες σχεδόν. Και αυτό που προτείνουμε είναι καταρχάς οι διατάξεις για τις εισερχόμενες κλήσεις, Δηλαδή θέλουμε να εξομαλύνουμε το καθεστώς περιαγωγής... Ε, όταν πρόκειται για εισερχόμενες κλήσει να είναι το φυσιολογικό. Στην Ευρώπη φυσιολογικά πληρώνει αυτός που τηλεφωνεί, όχι αυτός που δέχεται την κλήση. Και θέλουμε αυτό να ισχύσει και στην πυριαγωγή. Και από εκεί και πέρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα προαιρετικό καθεστώς, έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Με βάση την οπτική γωνία της αγοράς. Μπορούν οι παίκτες να κάνουν οικονομίες κλίμακας, ακόμα και αν δεν έχουν τέτοια δυνατότητα στο δικό τους δίκτυο, να έχουν ένα ευρωπαϊκό αποτύπωμα και να ε, προσφέρουν την περιαγωγή μέσω αμοιβαίων ε, συμφωνιών, οι οποίες ήδη υπάρχουν. Δεν επινοούμε δηλαδή την αγορά αυτή από το μηδέν, αλλά διασφαλίζουμε ότι αυτά τα ωφέλη θα μετακυλιστούν στους τελικούς χρήστες. Και αυτό άλλωστε είναι και δικό σας στόχος, όχι μόνο και δικό μας. Και, δικός μας. Ε, και μάλιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με δύο λόγια, απαντώντας στην κυρία Πάστος για το ότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε αλλάξει κάπως τη ρητορική μας, θέλω να πω το εξής. Με την πρόταση αυτή υπογραμμίζουμε την κλίμακα όχι ως ε, ουσία αυτή αυτή αλλά λέμε ότι η οικονομία κλίμακας που μπορεί κανείς να πετύχει, να μην φράσεται, να μην παρεμποδίζεται, να μην μπλοκάρεται από νομοθετικές διατάξεις σε όποιο πεδίο και αν αναφέρονται και σε όποιο πεδίο και αν ισχύουν αυτές οι διατάξεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ακόμα και όταν αναπτύσσουμε αναπτύσσονται οι εταιρείε και αυξάνουν το ευρωπαϊκό τους αποτύπωμα, δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί ο ανταγωνισμός και οι επιλογές που θα βιώσει ως εμπειρία ο τελικός χρήστης. Θέλουμε όλο και περισσότερο δυναμισμό της αγοράς και τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό επιλογών όσος είναι αυτός ο αριθμός επιλογών που έχει αυτή τη στιγμή ο τελικός χρήστης στην εθνική και τοπική του αγορά. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με όλα αυτά που κάνουμε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα να μην σπαταλίσω πολύ από το χρόνο της Επιτροπής σας. Νομίζω όμως ότι συνέβαλα στο να διευκρινιστούν κάποιες αμφιβολίες σας. Είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εμείς έχουμε καταχραστεί του χρόνου σας. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι η συζήτηση είναι δημόσια, γιατί παρακολουθούν οι άνθρωποι τη συζήτησή μας και μπορεί να υποβάλουν σχόλια. Εγώ άσκησα επικοδομητική κριτική της πρότασης αυτής. Έχουμε κάποια απογοητεύση. Πιστεύουμε ότι θα, είχαμε, θα είχατε καλύτερα ωφέλη, περισσότερα αποτελέσματα προς όφελος των καταναλωτών. Ίσως είναι λίγο αργά γι' αυτό. Και εγώ συμβουλεύτηκα τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και τους ζήτησα να μου πούν αν μπορούμε να υιοθετήσουμε τη μορφή αναθεώρησης της οδηγίας και μου είπαν ότι αν το είχαμε ξεκινήσει αυτό πριν από λίγους μήνες μπορεί και να πέρναγε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δικαίωμα ίδια πρωτοβουλία εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επελέξατε να μην ακολουθήσετε αυτή την άγουσα της αναθεώρησης οδηγίας. Ελπίζω να μην έχουμε χάσει κάτι με την ε, διαδρομή που έχουμε επιλέξει, που έχετε επιλέξει δεν μπορούν να γίνουν αλλαγέ στην νομική οδό που, θα, που έχει ήδη αποφασιστεί σε αυτό το στάδιο. Καλό ή κακό λοιπόν αυτή τη νομική οδό θα ακολουθήσουμε, αυτή που έχετε εσεί επιλέξει. Α ελπίσουμε ότι ε, θα κάνουμε το καλύτερο και θα δούμε και την συνεισφορά των κρατών μελών. Δεν θα υιοθετηθεί αυτή η δέσμη μέτρων και προτάσεων πριν από το φθινόπωρο του 2014 και μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέχρι τότε και ειδικότερα στην περιαγωγή πάρα πολλά πράγματα διασύνδεσης γίνονται. Άλλοι συνάδελφοι και πολλοί συνάδελφοι ε, ήδη έχουν ένα συμβόλαιο με συγκεκριμένο πάγιο και έχουν απεριόριστη περιαγωγή οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα αυτά είναι συμβόλαια που θα αρχίσουν να προτείνουν όλο και περισσότερε εταιρείε κινητή τηλεφωνία σε όλο και περισσότερου ανθρώπου. Σίγουρα θα γίνουμε μάρτυρε αναδιάρθρωση τη αγορά. Όλα αυτά είναι κοινοτομίε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τούτων λεχθέντων α περιμένουμε να δούμε. Ξέρουμε ότι όλοι θέλουν το καλύτερο για του καταναλωτέ Και είναι και το θέμα των περιορισμών στο voice over IP. Η ουδετερότητα είχε να κάνει με την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται, όχι με τη φραγή στην πρόσβαση στις υπηρεσίες. Και πρέπει να έχουμε εργαλεία πολύ υψηλής αξίας ως προς την προστασία του ανταγωνισμού και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των δικών μας υπηρεσιών, γιατί δεν είναι θέμα ποιότητας της υπηρεσίας, το, της ουδετερότητας. Και μία από τις διατάξεις που προτείναμε για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό είναι το εξής, ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει σαφέστατη προσυμβατική ενημέρωση για τις υπηρεσίες που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και δεν το έκαναν τόσο πολύ αυτό οι εταιρείε. Και θα πρέπει να έχουμε κανονισμούς ούτως ώστε να υπάρχει ένας τουλάχιστον πάροχος στην αγορά κάθε φορά που να είναι σε θέση να προσφέρει αυτή την εναλλακτική λύση. Απογοητεύομαι λοιπόν με τον τρόπο που ερμηνεύεται το επιχείρημα της ουδετερότητας, γιατί χρησιμοποιείται την ποιότητα, ε, το, γιατί χρησιμοποιείται η ποιότητα των υπηρεσιών για να υπάρχει διάκριση υπέρ του, των υπηρεσιών που προσφέρει μία εταιρεία σε σχέση με τις άλλες. Και δεν είναι αυτό η ουδετερότητα. Δηλαδή ο καθένας ερμηνεύει την ουδετερότητα διαφορετικά. Άρα καλώς τη βγάλατε την ουδετερότητα από τα σημεία που είναι προς συζήτηση. Το ότι τη βγάλατε όμως και καλώς δείχνει πόσο δύσκολη έννοια είναι και πόσο ρευστά είναι όλα τα πράγματα. Και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σε νομικό επίπεδο το να θεσπίζουμε νέες νομικές έννοιες για να προλάβουμε την έλευση νέων προβλημάτων είναι κάτι που δεν είχαμε ξανακάνει στην αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι και φιλοσοφικό κατά την άποψή μου το ερώτημα, ενδεχομένω οι συνάδελφοι διαφωνούν. Εν πάση περιπτώσει η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, αδειμονώ να συνεργαστώ με την κυρία Μπάστο, η οποία έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση αυτή τη πρόταση και οι άλλοι συνάδελφοί που θα συνεργαστούν μεταξύ του και σίγουρα θα οργανώσουμε ακρόαση όπου θα συζητηθούν αυτά τα θέματα ε, δημοσίω και θα ακούσουμε και από του νομοθέτε ε, ποια είναι η άποψή του για όλε αυτέ τι προτάσει, για το πώ εφαρμόζουν τι υφιστάμενε διατάξει που υιοθετήσαμε το 2009. Σα υπενθυμίζω επίση ότι δεν είναι ξένα για εμά τα ζητήματα τη εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών είχαμε μια μακροσκελή συζήτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις θελήσαμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερα ωφέλη στους καταναλωτές από ό,τι θα μπορούσαν να τους δώσουν με ένα εναρμονισμένο σύστημα. Το ίδιο πιστεύουν και πολλοί που στελεχώνουν το χώρο των τηλεπικοινωνιών. Είναι ένα πνεύμα, ένα κλίμα που έχει διαμορφωθεί εδώ Εν πάση περιπτώσει θα το προχωρήσουμε, θα τα προχωρήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που ήρθατε. Λυπούμε που δεν ήταν περισσότεροι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή, αλλά θα είναι ενδιαφέροντες οι τελευταίοι μήνες ε, που θα ασκήσω την Προεδρία σε αυτή την Επιτροπή, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε ενθουσιώδεις στη δική μας προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι είχατε την υπομονή να μας παρακολουθήσετε και να ξέρετε εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πολύ γρήγορα θα σας προσκαλέσουμε ξανά. Επόμενη συνεδρίαση την ε, Δευτέρα, λέει ο Πρόεδρος, 5 Νοεμβρίου, αλλά είναι 4 Νοεμβρίου τη Δευτέρα, από 3 μέχρι τις 6.30. Πενθήμερο στην Βρετανία και Τρίτη 6 Νοεμβρίου, λέει ο Πρόεδρος, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Θα τα πούμε τότε. Ευχαριστώ.